Colleagues. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την ε, μικρή καθυστέρηση. Είχα θέμα για να φτάσω από το ισόγειο στον τρίτο όροφο, γι' αυτό καθυστέρησα. Next item on the agenda. Λοιπόν, περνούμε στο σημείο 7 της μερίσιας διάταξης, ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις ε, αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύσκεψη των συντονιστών. Πρώτα απ' όλα έγινε μια παρουσίαση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από τον ΕΑΣΑ σε σχέση ε, με τη, τους, τις ώρες πτήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβαν γνώση οι συντονιστές των διαθέσιμων πληροφοριών και θα επανέλθουμε στο θέμα με το που αρχίσει και επίσημα η διαδικασία επιτροπολογίας. Σε σχέση με το διορισμό των εισηγητών, είχαμε κάποιες εκθέσεις πρωτοβουλίες για τις οποίες αποφασίσαμε. Πρώτον, ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την εξωτερική αεροναυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, μετά από ε, συμφωνήθηκε να ανατεθεί στο ΕΛΚ, στη συνέχεια έρευνα και κοινοτομία για την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά. Αποφασίστηκε να ανατεθεί στους πρασίνους. Κατόπιν ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μπλε αναπτυξιακό πολιτικό για την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι σοσιαλιστές ανέλαβαν το θέμα αυτό. Η απόφαση να μην αναλάβουμε δράση ε, σε σχέση με τα συστήματα αεροπλοήγησης, τι λέει συστήματα αεροπλοήγησης, ε, καθώς και για την εφαρμογή ε, των ηλεκτρονικών τελωνίων, ε, διοδίων, συγγνώμη, ανατέθηκε στο ΕΛΚ. Έγγραφα που λέγαμε προς ενημέρωση, ε, ε, γνωμοδοτήσεις για την απαλλαγή 2011 για το σύστημα εκπεριτροπής. Οι πράσινοι θα αναλάβουν την ε, απαλλαγή του 2011 για τον συνολικό προϋπολογισμό της ευρωπαϊκή Ένωσης και οι φιλελεύθεροι θα ασχοληθούν με την ε, απαλλαγή για τους τέσσερις, για, τους οργανισμούς που μας απασχόλησαν. Σε σχέση τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου ε, για ε, τα συνδεδεμένα εδάφη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, δεν αποφασίστηκε τίποτα, ούτε και αποφασίστηκε τίποτα σε σχέση με τις διατάξεις για το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν κάνουμε τίποτα για τον πίνακα απλούστευσης, ούτε και για το έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές. Στη συνέχεια προτάθηκε να ανανεωθεί το σύστημα βαθμών ε, αυξάνοντας ε, τον βαθμό αναλογικά με τον αριθμό των μελών της κάθε πολιτικής ομάδας ε, και οι τέσσερις ομάδες διαφωνούσαν για... Έχουν ένα βαθμό επικαιροποιούμε το σύστημα βαθμών λοιπόν και αυξάνουμε το, τον αριθμό των βαθμών αναλογικά με τον ε, αριθμό των μελών της κάθε πολιτικής ομάδας. Καταψήφισαν οι πράσινοι την πρόταση. Ένα λεπτάκι θα σας δώσω το λόγο. Καταψήφισαν λοιπόν την πρόταση οι πράσινοι εξετάσαμε και έναν άλλο τρόπο κατανομής των βαθμών που εισηγήθηκαν εξάλλου οι πράσινοι. Οι συντονιστές όμως αποφάσισαν να παραμείνουν ε, στο ε, ισχύον σύστημα. Η συμφωνία δεύτερη ανάγνωση για του ταχυγράφου συμφωνήθηκε ο εισηγητή να ε, λάβει την εντολή για να αρχίσει διαπραγματεύσει με την Κυπριακή Προεδρία επί τη βάση του αποτελεσμού της πρώτης ανάγνωσης και με την πλήρη συμμετοχή των σκιωδών εισηγητών. Ε, το ενημερωτικό δελτίο για την επιτροπολογία επίσης ε, κυκλοφόρηση για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας TNT. Ε, λάβαμε μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και καταγράψαμε τις πληροφορίε που μας έδωσαν οι πρόσωποι τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα διαφορά. Ε, μία επιστολή προς την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών σε σχέση με το ρόλο που θα έχουν το 2030 τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, η επιστολή βασίζεται ε, στο σύστημα της στενής συνεργασίας των εισηγητών με τους αντίστοιχους εισηγητές από τα Εθνικά Κοινοβούλια κατά την κατάσταση των γονομοδοτήσεων. Ε, στη συνέχεια, εξωτερική τεχνογνωσία και τα σχετικά προγράμματα συμφώνησαν οι συντονιστές να ζητήσουν ένα πρόγραμμα για ε, τα Giga Lines, τα μεγάλα και βαρέα φορτηγά κατά το δεύτερο κύκλο του προϋπολογισμού και να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα για όλα τα σχέδια του 2013. Μελέτε δηλαδή είναι και σε σχέση με τι τεχνικέ εξελίξει. Ε, και την εφαρμογή για την καταγραφή των δεδομένων στον τομέα τη οδική ασφάλεια. Ε, ζητήθηκε ανάλυση σε σχέση με τι τεχνικέ εξελίξει ε, και την υλοποίηση χρήση νέων συσκευών στον τομέα των οδικών μεταφορών καθώ και εξέταση του σημείου των οδικών μεταφορών σε απομακρυσμένε περιοχέ. Στην επόμενη συνεδρία τη επιτροπή οι συντονιστές θα εξετάσουν μια άλλη συζήτηση σε σχέση με την επανακατάρτιση τη πρόταση. Ε, για το πακέτο ε, για τις αεροπορικές ε, μεταφορές και θα διοργανωθεί, διοργανωθεί συνεδρίαση με το που βρούμε αίθουσα και χρόνο. Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Κάποιοι συντονιστέ και κάποιοι εισηγητέ δεν μπορούσαν να παρευρεθούν και δεν καταλήξαμε συμφωνία. Προτάθηκε λοιπόν ανταυτού μετά από πρωτοβουλία του ΕΛΚ ε, να ε, μετατεθεί το θέμα ε, στις 6 Οκτωβρίου, στις 3, δηλαδή θα ψηφίσουμε για το πακέτο των αερομεταφορών. Θα αρχίσει η ψηφοφορία στις 3 το απόγευμα στις 6 Οκτωβρίου και όλα τα υπόλοιπα που είχαν προβλεφθεί για το απόγευμα θα μεταφερθούν το ίδιο πρωί, ούτως ώστε να έχουμε μισή μέρα με τρόπο ώστε οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές να έχουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να καταλήξουν συμβαστικέ λύσεις ή στην γενικό γενικότερη δομή των εργασιών μας, ε, διότι έχουμε εκατοντάδες τροπολογίες, ε, χιλιάδες ε, τροπολογίες για το πακέτο των αεροπορικών μεταφορών και δεν είναι το μόνο ζήτημα. Δεν ξέρω ε, πόσο δυνατοί είσαστε, αλλά ούτε εγώ δεν θα μπορούσα ε, να το κάνω παρά την ταχύτητά μου και ε, κρίναμε ότι η καλύτερη λύση ήταν ε, να μην διοργανώσουμε νέα συνεδρία, απλώς να μεταφέρουμε το θέμα το απόγευμα εκείνη τη ημέρα, 6 Οκτωβρίου, όπως σας εξήγησα. Κραμ και Λάιφριντ, Παρακαλώ. Είπατε ότι είμαστε αντίθετοι με το σύστημα των βαθμών ή των πόντων. Θέλω να επεκταθώ. Πρώτον, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα, είπαμε, αλλάζει όμως. Ε, επαναλαμβάνουμε αυτά που κάνει ο Κάλλας με το Liners, ε, με τα φορτηγά, δεν αλλάζω τους νόμους, αλλάζω την ερμηνεία τους. Τι λέει ο κανονισμός όταν τελειώσουν όλοι οι πόντοι και οι βαθμοί και έχουν μηδενιστεί όλα τα κοντέρ, τότε παίρνουμε και άλλους πόντους με βάση το σύστημα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική ομάδα που να είναι στο μηδέν, αλλά το αλλάζεται επειδή τέσσερις ε, ομάδες έχουν ένα βαθμό, το αυξάνεται και αυτό στρέφεται κατά των μικρών ομάδων, δηλαδή ημών. Να το κοιτάξει η γραμματεία, είναι αλλαγή κανονισμού αυτό ε, ο κανονισμός ισχύει για το σύνολο τη θητείας. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε επειδή έτσι ταιριάζει ε, σε Ορισμένε ομάδε και ο Ματιό Γκρό είπε «Μα για εμά είναι ευνοϊκό, γιατί να είμαι αντίθετο. Ε, για εμά είναι δυσμενέ και είμαστε αντίθετοι. Τι του κάνουμε του κανόνε, ισχύουν για όλη τη θητεία. Δεν του αλλάζουμε όπω μα καπνίζει επειδή βολεύει κάποια πολιτική ομάδα και κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ να το εξετάσει η γραμματεία και επιφυλασσόμεθα κάθε δικαιώματό μα. Ε, το λέει σαφώ ο κανονισμό αυτό το πράγμα. Ε, νέους βαθμούς, ε, ίσως με τον αριθμό των μελών, θα λαμβάνουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή οι πέντε πολιτικές ομάδες έχουν εξαντλήσει τους πόντους και θα έρθουν να προσθεθούν. Ε, αλλά μέχρι τώρα καμία ομάδα δεν έχει φτάσει στο μηδέν. Γιατί να αλλάξουμε το σύστημα, ή το. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Okay, well, actually, there are no formal rules about... Μάλιστα δεν υπάρχουν ουσιαστικά επίσημοι κανόνε για την κατανομή των βαθμών ε, Μάικλ. Κάθε επιτροπή ε, δράκατα το δοκούν και σε βάση περιπτώσει εναπόκειται στην ε, ευχαίρεια των συντονιστών. Εκείνοι το αποφασίζουν και στην αρχή είχαμε πει, δεν είχαμε πει για μηδέν βαθμού για τι πέντε ομάδε. Αν θυμάστε μιλήσαμε για την εξή πρόταση. Πρώτον πρόταση των φιλελευθέρων να τροποποιηθεί το σύστημα και τρει ή τέσσερι ομάδες να έχουν ένα αυτή είναι η ανακατανομή που γίνεται αφού λάβουν από ένα βαθμό και οι συντονιστέ τη Επιτροπή μα το αποφάσισαν και ξαναλέω, ε, ε, εργάζονται με διαφορετικό τρόπο. Ε, οι επιτροπέ γνωρίζουμε ότι προβάλλουν ένσταση οι πράσινοι, αλλά εν τέλει σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε, επικρατεί η πλειοψηφία. Αυτά μας είπαν όταν ήρθαμε σε επαφή με την ΑΦΚΟ και η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται, διότι οι τρεις πολιτικές ομάδες είπαν ότι θέλουν να ε, τροποποιήσουν το σύστημα κατανομής και να αλλάξουμε τους κανονες τοσο ούτως ώστε τρεις-τέσσερις ομάδες να έχουν ένα βαθμό και στη συνέχεια θα κάνουμε ανακατανομή. Έχουμε βρεθεί σε αυτό το στάδιο λοιπόν της ανακατανομής και προτείνουμε να ανανεώσουμε, να τροποποιήσουμε το σύστημα. Μπορούμε να κάνουμε μια επίσημη ψηφοφορία, αλλά είναι λίγο άσκοπο κατά τη γνώμη μου, γιατί θα έχουμε συντριπτική πλειοψηφία υπέρ αυτή τη πρόταση. Ε, καταγράφω τη διαμαρτυρία σα ε, και την ψήφο κατά τη πρόταση, αλλά μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση για την αύξηση των βαθμών επί του συστήματο που μόλι σα εξήγησα. Ε, γι' αυτό το θέμα, κυρία Μάιστερ. Ναι, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό, γιατί εχθέ αποσίαζα. Ήθελα να πω ξανά ότι εγώ το πρότεινα, παρόλο που είναι δυσμενέ για μας και εγώ ε, δεν είμαι από μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά δεν υπάρχει ομάδα που ε, θέλει να δαπανίσει τώρα ένα ε, θέμα πολύ σημαντικό που είναι το road charge system ε, και γιατί δεν θέλει να χάσει αυτό το βαθμό τη. Γι' αυτό λέω να έχουμε περισσότερους πόντους για να μπορούμε να του ξοδεύουμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Γι' αυτό το πρότεινα. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο πολιτικές ομάδες που δεν παίρνουν ποτέ έκθεση, παρόλο που έχουν δύο πόντους. Και αυτό είναι πολύ ατυχές. Δεν πρόκειται ποτέ να μηδενίσουν αφού δεν παίρνουν ποτέ έκθεση. Α, και ένα τελευταίο. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά και αυτό το point system που έχουμε είναι πάντα η πέτρα του σκανδάλου. Ε, δεν μπορούμε να δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε έτσι αρμονικά. Θέλω να επανέλθει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ό,τι και να γίνει στη νέα θητεία, τότε θα είναι η σωστή στιγμή για να εξετάσουμε και να μιλήσουμε για το σύστημα βαθμών που επιθυμείτε. Το η δουλειά των συντονιστών είναι να εφαρμόσετε σωστά το σύστημα. Ο κύριος Κράμερ, θέλω να επαναλάβω ότι εντάξει, στι διάφορε επιτροπέ ισχύουν διαφορετικοί κανόνε, αλλά αυτή τη στιγμή βάζει κανόνε, αυτοί ισχύουν για το σύνολο τη θητεία και δεν μπορούν να αλλάξουν. Το γνωρίζω το πρόβλημα. Αλλά αυτό έχει διεκπεριωθεί, γιατί στην παρούσα θητεία δεν θα έχουμε πια εμείς την ευκαιρία να πάρουμε έκθεση, θα το κάνουμε δύο μεγάλες ομάδες και εντάξει, θα επανέλθει τάξη και ασφάλεια και ησυχία. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να πάρουμε έκθεση. Ε, κοιτάξτε, ξαναλέω ότι η Επιτροπή κάνει ό,τι θέλει με το δικό της σύστημα κατανομής. Μάικλ, αυτό είναι ένα ε, δεδομένο. Προτείνω να ε, λήξει η συζήτηση. Κύριε Λάιχφριντ, για κάτι άλλο ζητήσατε το λόγο, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Μια ερώτηση έχω. Το πακέτο των αεροδρομίων δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το απόγευμα. Γιατί με τις τροπολογίες μπορεί λίγο να μπλέξουμε, ε, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν γνωρίζω αν ισχύει, αλλά κατά την άποψή μου ε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την Τρίτη πριν την ψηφοφορία της τροπολογίας. Γιατί αυτό μας δίνει ένα περιθώριο χρόνου. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα βέβαια να αλλάξουμε τώρα ε, την ημερήσια διάταξη. αν θέλετε να εξεταστούν το πρωί οι τροπολογίες και το απόγευμα να ψηφίσουμε, εντάξει, τέλος πάντων, αν χρειαστούν προσαρμογές δηλαδή. Εγώ αυτό που εννοούσα είναι ότι είναι μάλλον καλύτερα να γίνει αυτό τη Δευτέρα και όχι την Τρίτη. Αλλά, αλλά εσείς αποφασίζετε για αυτό το θέμα. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι η ψηφοφορία. Νομίζω μόνο η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει τόσο σε περιόδους ψηφοφορίας. Εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τον επιπρόσθετο χρόνο για να μπορούμε να συζητήσουμε το απόγευμα. Και συνεχίζω να ελπίζω ότι με τη μεταφορά στο απόγευμα θα λειτουργήσουν όλα πιο εύρυθμα. Ίσως να ασφάλω κιόλας, αλλά... Θα δούμε, αλλά θα πρέπει να διαβολευτούμε με τους συντονιστές αν θεωρούν ότι είναι καλύτερο να γίνει συζήτηση την ίδια μέρα το πρωί, ας το κάνουμε, αλλιώς θα αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Συμφωνείτε με αυτό, κύριε Κράμερ? Μα, είχε γίνει μια πρόταση να αναβληθεί η ψηφοφορία για τις 12 Νοεμβρίου. Τι έγινε, αυτό καταργήθηκε, δεν γίνεται, δεν το έχετε εξτάσει. Μάικλ, όταν ε, εισήγαγα το σημείο, ανέφερα τα προβλήματα για τη 12η Οκτωβρίου, διότι δεν μπορούν να... Ε, την, ε, για 12η Νοεμβρίου δεν μπορούν να έρθουν οι συντονιστές, δεν μπορούν να έρθουν οι συγητές και εγώ ίδιος δυσκολεύομαι. Προσπαθήσαμε λοιπόν να υπερπηδήσουμε αυτό το εμπόδιο και προτάθηκε να μετατεθεί η νοεμβριου δεν μπορουν να ερθουν οι συντονιστες δεν μπορουν να ερθουν οι συγητες και εγω ιδιος δυσκολευομαι προσπαθησαμε λοιπον να υπερβιδισουμε αυτο το εμποδιο και προταθηκε να μετατεθει η ψηφοφορια στις 12. Είναι το εφεδρικό σχέδιο και θυμάστε ότι στους συντονιστές ε, το συμφωνήσαμε να κάνουμε την ψηφοφορία το απόγευμα στις 6 Οκτωβρίου. 6 Νοεμβρίου. Η πράσινη είναι κατά της, ε, της πρώτας ανακατανομής ε, των βαθμών. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν. Ε, Λίγοι και αυτό το σημείο. Επόμενο. Η ειδική ομάδα για τον τουρισμό του κυρίου Φιντάνση. Ε, η ομάδα αυτή τον Ιούλιο συνεδρίασε και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις μη προτεραιότητες της ομάδας για τους προσεχείς μήνες. Θα θυμάστε ότι συστάθηκε αυτή η ειδική ομάδα μετά από ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ε, ζητήσαμε από τον κύριο Φιντάνζε να συντάξει αυτό το κείμενο για να συλλέξει και παρατηρήσεις και σχόλες. αυτό το στάδιο θα του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει το έγγραφο αυτό. Να, να Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχετε πάρει από χτες αυτό το σχέδιο εγγράφου εργασία και ζητώ συγγνώμη εξ αρχής γιατί για λόγους χρόνου ε, δεν μπόρεσα να σας στείλω και τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες. Ε, γι' αυτό πήρατε μόνο μία εκδοχή στα αγγλικά. Ε, αυτό βέβαια με περιορίζει, με υποχρεώνει να σας το εξηγήσω το κείμενό μου, ακόμα και αν το κάνω σύντομα. Να σας ε, πω κάτι για τη μεθοδολογία. Όπως είπαμε στην συντακτική συνεδρίαση της Task Force, αυτό το έγγραφο εργασίας είναι όντως έγγραφο εργασίας. Δεν είναι μια δεύτερη έκθεση, όπου, ένα κείμενο δηλαδή όπου επανεισάγουμε όλα όσα είχαμε βάλει στην ε, έκθεσή μας. Είναι ένα έγγραφο εργασίας, επί τη βάση του οποίου εντοπίζουμε ε, κάποιες προτεραιότητες και κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να προωθηθούν με, με βάση αυτές τις προτεραιότητες. Είναι βασικό λοιπόν, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτό το έγγραφο και να μιλήσουμε και για προτάσεις ολοκλήρωσης σε αυτό το πνεύμα. Δηλαδή να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και σε, με βάση, μάλλον με στόχο συγκεκριμένες προτάσεις από πλευράς μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους που έχουν ήδη στείλει σχόλια. Κάποια από αυτά τα έχω ήδη συμπεριλάβει στη σημερινή εκδοχή του κειμένου. Έχουμε επίσης εδώ ε, υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, του Τμήματο για τον Τουρισμό. Θα έχουμε δηλαδή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει μαζί του. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας αναφέρω όλα τα σημεία. Καταρχήν, έχω προτείνει να χωριστεί αυτό το έγγραφο εργασίας σε πέντε τομείς προτεραιότητας. Ο πρώτος είναι η προώθηση της συνεργασίας, δηλαδή χρειαζόμαστε, όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει στα έγγραφα που έχουμε ψηφίσει και στις συζητήσεις μας, χρειάζεται ο οριζόντιος χαρακτήρας των πολιτικών του τουρισμού και το διαφορετικό επίπεδο αρμοδιοτήτων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, να μας οδηγήσουν στο να αυξήσουμε το επίπεδο της ε, διαθεσμικής συνεργασίας. Γι' αυτό οι συγκεκριμένες προτάσεις που προκύπτουν από αυτήν ε, την ε, σκέψη είναι να βάλουμε εξ αρχής από την, από την επόμενη σύνοδο της Επιτροπής μας ε, να, να, να, διοργανώσουμε μια συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Αρμόδιο για τον τουρισμό κύριο Ταγιάννη και μετά θα πρέπει να αξιολογήσουμε και γι' αυτό εγώ είμαι ανοιχτή, ανοιχτός μήπως ε, θα πρέπει να κάνουμε και μια συνάντηση με την Κυπριακή Προεδρία αν και βέβαια ε, θα έχουμε πια προχωρήσει προς το τέλος αυτής της ε, Προεδρίας ή μήπως θα είναι καλύτερα να διοργανώσουμε για τον Ιανουάριο ε, μία επαφή με τον Υπουργό Τουρισμού της επόμενης Προεδρίας που θα ξεκινήσει με τον καινούριο χρόνο. Επίσης, μέσα στις επαφές που θα μπορούσαμε να έχουμε παράλληλα με τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, που κατά προτεραιότητα ενδιαφέρονται για τα θέματα τουρισμού. Να έχουμε λοιπόν από εκείνες μια παρουσίαση της κατάστασης προόδου σε σχέση με τις δικές τους δραστηριότητες. Γιατί η ιδέα μου, η προσωπική, είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα, ε, να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να μην ε, αναλαμβάνονται θεωρητικές συζητήσεις σε σχέση με δράσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η Κομισιόν και μάλιστα σε μερικέ περιπτώσει μετά από υποδείξει του Κοινοβουλίου. Να δούμε δηλαδή από τι γενικέ διευθύνσει τη Κομισιόν τι κάνουν πραγματικά, ώστε να αποφύγουμε επικαλύψει και να μην χάνουμε χρόνο σε θεωρητικέ συζητήσει σε σχέση με θέματα που ήδη αντιμετωπίζονται στην πράξη. Επίσης, μια μεθοδολογική πτυχή που απορρέει από τις προτεραιότητες που θα εγκρίνουμε με αυτό το έγγραφο εργασία είναι παράλληλα με τις επίσημες ε, συνεδριάσεις που έχουμε εδώ να διοργανώνουμε και επαφές και θεματικές συνεδριάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Ε, κάτι ακόμα αφορά τη συνεργασία με τις άλλες επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου. Το έχουμε συζητήσει αυτό στην συντακτική συνεδρίαση της Task Force. Ακριβώς λόγω της ε, οριζόντιας του φύσης, ο τουρισμός έχει φυσικά αντίκτυπο σε αποφάσεις για ρυθμίσεις ή κανονισμούς που αναλύονται και υπερψηφίζονται από άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρέπει να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι προτεραιότητες που αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση στις υπόλοιπες επιτροπές του Κοινοβουλίου, να διοργανώσουμε διμερείς επαφές με αυτές τις επιτροπές, ώστε να εξηγήσουμε τις απόψεις και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ορισμένες αποφάσεις στον τουρισμό. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μεταξύ άλλων ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση στην Επιτροπή Ήτρε για το πρόγραμμα COSME, για τη στήριξη δηλαδή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ξέρετε ότι εκεί περιλαμβάνεται ένα σημαντικό κονδύλι για τη στήριξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό που θα πρέπει να την υπερασπίσουμε. Και έχουμε ήδη ψηφίσει εξάλλου μια γνωμοδότηση δική μας για το πολιετές ε, πλαίσιο, στηρίζοντας ε, το ότι χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένη γραμμή για τον τουρισμό. Έπειτα, ε, δεύτερη προτεραιότητα, η προώθηση του τουρισμού για όλους. Εδώ έχω χωρίσει αυτό το μεγάλο θέμα σε δύο υποπροτεραιότητες. Η μία είναι η προσβασιμότητα και η δεύτερη εποχικότητα. Για την προσβασιμότητα, δυνατότητα πρόσβασης, έχουμε ήδη συζητήσει, έχουμε διοργανώσει και ακροάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο διαρκώς ανεβαίνει στην ε, κοινή γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς δεσμεύεται και περισσότερο και πιστεύω πως επ' αυτού το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει καλή δουλειά και έχω μάλιστα λάβει και διάφορα αιτήματα από πλευρά των συναδέλφων. Και το μέγα θέμα της εποχικότητας, το οποίο μπορέσαμε επίσης να δούμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και όσοι μαζί μας ήρθαν στην Κρήτη, σε όλες τις επαφές που είχαμε, είδαμε ότι είναι ένα από τα βασικά επίγοντα θέματα των τουριστικών μονάδων. Δεν μπορούν να επιβιώσουν ε, ε, δουλεύοντας ένα-ενάμιση ένα, μήνα, άντε δύο το χρόνο. Πρέπει δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε αυτή την άκομπτη εποχικότητα του τουρισμού επίσης επαφές με την Κομισιόν ώστε να εντοπίσουμε δράσεις που μπορούν να συνεχιστούν με βάση τα όσα έχει γίνει στο παρελθόν, όπως ας πούμε το καλυψό να βρούμε τι θα κάνουμε μετά από το καλυψό που τελειώνει εκπνέει φέτος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την εποχικότητα. Αυτές οι δύο πτυχές συνδέονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό και εγώ ανέκαθεν έλεγα ότι η εποχικότητα ξεπερνιέται μέσω της δυνατότητας ε, των λιγότερο προνομιούχων κατηγοριών πολιτών να μπορούν να ταξιδεύουν σε, στις χαμηλές περιόδους. Θα μπορούσαμε δηλαδή να βρούμε συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξουμε εδώ την κατάσταση. Ορισμένοι συνάδελφοι πρότειναν να μείνουν αυτά χωριστά. Θα δούμε, θα το δούμε. Εγώ είμαι ανοιχτό αυτό πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού. Το μόνο θέμα είναι να αποφύγουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Θα το δούμε λοιπόν με τον Πρόεδρο. Ίσως θα ήταν καλύτερο να εστιάσουμε την προσοχή σε ένα από όλα. Μας περιπτώσει θα το δούμε αυτό μαζί, θα το αξιολογήσουμε. Τρίτη προτεραιότητα, στήριξη στη διαφοροποίηση της ε, τουριστικής προσφοράς. Πρέπει να έχουμε υπόψη το, το γεγονός ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πολυάριθμες ε, τουριστικές ε, ε, τουριστικούς προορισμούς, τόσο όσον αφορά τα διαδρομές, τόσο όσον αφορά και την τυπολογία της, των προορισμών αυτών, θα πρέπει αυτό να το θεωρήσουμε ως προσθέμενη αξία εν γέννη και να διατηρήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση καθώς και να δουλέψουμε με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη ε, διαφοροποίηση για να στηρίξουμε τις διαδρομές αυτές που υπάρχουν ε, και αυτές που μπορούν να δημιουργηθούν. Υπάρχουν ένα σωρό πολιτιστικές, ε, πολιτιστικές διαδρομές, φυσιολατρικές διαδρομές και ούτω καθεξής, αλλά μπορούμε να προωθήσουμε και συγκεκριμένους τομείς, όπως πούμε ο επαγγελματικό τουρισμός, ο επαγγελματικό συνεδρίων, ο, ο τουρισμός Τη της Υπέθρου. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και στο δεύτερο πυλώνα υπάρχει το θέμα της ανάπτυξης της Υπέθρου σε σχέση με τον τουρισμό. Μια ολόκληρη σειρά δηλαδή εδώ συμβολών που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τέταρτη προτεραιότητα, η προσέλκυση νέων ροών. Και εδώ υποδιαιρώ το θέμα σε δύο υποπροτεραιότητες. Το πρώτο αφορά την πολιτική θεωρήσεων, γιατί τακτικά έχουμε στηρίξει και έχουμε διαπιστώσει πως μια πολιτική θεωρήσεων σε ορισμένε περιπτώσεις είναι εξαιρετικά περιοριστική, πράγμα το οποίο επιφέρει ανταγωνιστικό μεονέκτημα στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημιουργείται και διαφορά, υπάρχει μάλλον διαφορά ανάμεσα στις χώρες σε σχέση με τις διαδικασίες, το χρόνο που παίρνουν αυτές, ε, το κόστος τους, ε, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό από πέρσι εμείς στηρίξαμε το ότι χρειάζεται μια εναρμόνιση στις ε, διαδικασίες ε, χορήγησης ε, θεωρήσεων και απλοποίηση προς τις χώρες BRIC που μπορούν να δώσουν στην Ευρώπη μια νέα και μεγαλύτερη ροή δυνητικών τουριστών. Γι' αυτό και έχετε την πρόταση στο έγγραφο εργασίας εδώ Καταρχήν να έχουμε πρώτα μια επαφή με τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης της ε, Ένωσης και ευχαριστώ τον συνάδελφο Δανέλη για αυτή την πρόταση και έπειτα να κάνουμε και μια προφορική ερώτηση με συζήτηση στην Ολομέλεια για την πολιτική θεωρήσεων στην Ευρώπη που όπως γνωρίζετε είναι μια αρμοδιότητα την οποία έχει η Επίτροπος Μάλστρομ αν δεν κάνω λάθος και έτσι Δευτερευόντως ε, ασχολείται και ο Επίτροπος ε, Ταγιάννη που είναι απέθυνος για τον τουρισμό ε, αλλά και να δούμε και τις εσωτερικές υποθέσεις, δηλαδή τη ρύθμιση για τη, τις ρυθμίσεις για τη μετανάστευση και το καθεξής. Αφορά δηλαδή όλο το κοινοβούλιο αυτό το θέμα και όχι μόνο εμάς. Έπειτα, δεύτερη άλλη προτεραιότητα, η πρόθεση της Ευρώπης ως ποιοτικής, ποιοτικού μάλλον τουριστικού προορισμού. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε εντάξει στην εργασία μας εδώ στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα το θέμα της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Σήματος, European Brand. Άλλη προτε... πέμπτη προτεραιότητα, επένδυση στην ποιότητα. Εμείς έχουμε επανειλημμένω επιβεβαιώσει ότι η ποιότητα μαζί με τη διαφοροποίηση τη προσφορά είναι μια από τι προστιθέμενες αξίε τη Ευρωπαϊκή Τουριστική προσφορά σε σχέση με άλλους ε, τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Επ' αυτού εγώ έχω εντοπίσει δύο κύρια θέματα. Το πρώτο είναι η ετικέτα και έπειτα το σύστημα ε, ταξινόμησης. Είναι δύο θέματα ε, πολύ επίμαχα για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας. Η Κομισιόν έχει ήδη δεσμευτεί εδώ και μήνες για μια σειρά δράσεων. Έχουν γίνει ε, συζητήσεις, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν ορισμό ενός κοινού σήματος όπου προβλέπει μίνιμουμ ε, προδιαγραφές ποιότητας αναγνωρισμένων ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια, ένα γενικό σήμα, ομπρέλα, στο οποίο θα μπορούν να προσχωρήσουν τα διάφορα σήματα ποιότητας που ήδη υπάρχουν στα διάφορα κράτη. Εγώ μπόρεσα να συμμετέχω ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου σε κάποιες από αυτές τις ε, συναντήσεις. Εγώ πιστεύω πως δεν χρειάζεται να κάνουμε πάλι αυτή τη δουλειά που κάνει ήδη η Κομισιόν με διάφορους φορείς, γιατί σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε πολλές συνεδρίες γιατί δεν βρίσκουμε άκρη. Πάντως, είναι σημαντικό να γίνει μια επαφή με τους απεύθυνου για αυτά τα θέματα της Κομισιόν για να καταλάβουμε πού καταλήγουν εκείνοι και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως Κοινοβούλιο. Άλλο ε, καθόδες θέμα είναι το σύστημα το... της ταξινόμησης των ξενοδοχείων. Μιλώντας στα Σανσέρ, είπαμε και συμφωνούμε όλοι ότι στην Ευρώπη του 2013 επικρατεί ένα σύστημα με αστέρια που δεν είναι ομοιόμορφο για όλες τις χώρες και πολλές φορές και μέσα στην ίδια χώρα δεν είναι το ίδιο ένα τετράστερο ξενοδοχείο στο Μπολτζάνο με ένα τετράστερο της Λαμπεντούζα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές που που οδηγούν σε σύγχυση και αβεβαιότητα σε σχέση με την προσφορά που θα βρει ο, ο τουρίστας. Η πρόταση που κάνω, φοβάμαι πως ούτε η επόμενη θητεία δεν θα αρκέσει για να φτάσουμε σε συγκεκριμένη λύση, ούτε και η μεθεπόμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει ως κοινοβούλιο να προωθήσουμε την εξέβρεση, την αναζήτηση τουλάχιστον μιας λύσης. Έπειτα, απαντήσεις ε, υπογραμμίσαμε εδώ, μάλλον και δράσεις, πως ο τουρισμός βασίζεται σε πόρους που εμείς α, χορηγούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση από τα διαρθρωτικά ταμεία και μετά εξαρτάται από τις ε, τοπικές και εθνικές αρχές πώς θα τα κατανείμουν αυτά στις περιφέρειές τους. Εν τω μεταξύ, Είδαμε όμως ότι στην πράξη συχνά αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή ε, κονδύλια τα οποία θεωρητικά απευθύνονται στον τουρισμό συχνά χρησιμοποιούνται είτε για να γίνουν εκστρατείε ε, προώθηση που δεν είναι καν καλές είτε για θέματα τα οποία τύπη είναι μόνο για τον τουρισμό, ενώ τελικά εξυπηρετούν τη χρηματοδότηση τοπικών μέτρων, μικρών υποδομών μεταφορών και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να είναι καρποφόρα τα χρήματα που ήδη υπάρχουν και που συχνά είναι κρυμμένα μέσα σε κεφάλαια δαπανών που δεν απευθύνονται ρητά στον τουρισμό. Η δεύτερη πτυχή είναι η πτυχή των πόρων που άμεσα δίνονται για τον τουρισμό ε, και έτσι επανέλθουμε στα αυτά που έλεγα αρχικά, ότι δηλαδή να ξεκινώντας με το πρόγραμμα COSME, για να προβλέψουμε για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης που μας αναθέτει την αρμοδιότητα για τον τουρισμό, την ε, πρόβλεψη ενός, ε, μιας γραμμής του προπολογισμού συγκεκριμένη για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων τουρισμού. Τελειώνω, Πρόεδρε στο τελευταίο κομμάτι του κειμένου θα δείτε και άλλα τρία θέματα που είναι κεντρικά και τα οποία έχουμε εντοπίσει εμείς στην έκθεσή μας και που είναι το θέμα της ε, επαγγελματική κατάρτισης, το θέμα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στον τουρισμό και το θέμα της ε, βιωσιμότητας, δηλαδή κλιματικές αλλαγές, πολιτική τουρισμού που να προσέχει περισσότερο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτά τα τρία θέματα ήθελα να τα αφήσω ανοιχτά, γιατί βρήκα κάποια δυσκολία στο να εντοπίσω συγκεκριμένε δράσει που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε για τα θέματα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το τεχνέ τεχνολογίε, γιατί υπάρχει ήδη μια τράπεζα εργασία που έχει φτιάξει η Κομισιόν με του βασικού ε, ενδιαφερόμενου φορεί του τομέα και δουλεύουν πριν να προβλέψουμε εμεί δε ε, δράσεις θα ήταν καλό ίσως να δούμε με την Κομισιόν πού βρίσκονται εκείνοι σε αυτή τη δουλειά για το θέμα της βιωσιμότητας και το θέμα των νέων τεχνολογιών, ώστε να καταλάβουμε ποιες προτάσεις μπορούμε συγκεκριμένα να ε, θέσουμε, να, υποβάλουμε. Να τελειώσω λέγοντα το εξή, ότι σίγουρα αυτό το κείμενο παραμένει ανοιχτό. Περιμένω και περαιτέρω δικά σα σχόλια, αφού θα έχετε λάβει την μετάφραση, γιατί ε, συνειδητοποιώ ότι ίσω να μην μπορούν όλοι να το δουλέψουν το κείμενο στα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένω δικά σας σχόλια ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε τη δημιουργία κάποιων ε, θεματικών ομάδων εργασίας για να απτύξουμε αυτές τις προτεραιότητες και να δώσουμε συνέχεια στις δράσεις που έχουμε αποφασίσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φιντάνσα. Έξι ομιλητές έχουμε προς το παρόν. Αν θέλετε και αλλάξετε γνώμη και θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε να μας το πείτε και θα δούμε πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Yes, Mr. Kramer, Mr. Perker, Mr. Higgins. Okay, put Mrs. Estras on and put your number one, Mr. Κυρία Βλάστο, πρώτη πρώτη είστε. To those seven speakers, and then we'll hear from Mr. Uh, Mr. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον κύριο Όρτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτό το πρώτο γύρο. Δύο λεπτά έκαστος ε, για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Ξέρω ότι χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο για να σας πω τα περί συντονιστών. Κυρία Βλαστού, σας παρακαλώ να τηρήσετε αυτά τα δύο λεπτά. Θα είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε ο συνάδελφος, ε, ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και βλέπουμε σήμερα ότι τονίζεται και η σημασία του ζητήματος. Ε, χάρη σε αυτό το έγγραφο, η ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού είναι μια πραγματικότητα πλέον για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ε, διότι αυτός ε, ο τομέας είναι σημαντικό, σημαντική συνιστόσα της οικονομίας μας και είναι και ένα φυτόριο θέσεων απασχόλησης πολύ σημαντικό δεδομένης της σημερινής κατάστασης. Μιλάμε για διάφορε πρωτοβουλίε ε, για τι οποίε πρέπει να βρούμε και την επαρκή χρηματοδότηση, χάρη στι οποίες, όπως μας είπε ο συνάδελφος, μπορούμε να προβάλλουμε ε, τα πλεονεκτήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να προαγάγουμε το ευρωπαϊκό σήμα, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρόκειται για να είναι ένας πλούσιος ταξιδιωτικός προορισμός. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διάφορα είδη τουρισμού, διάφορες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υποφεληθούμε από αυτό για να προσελκύσουμε τουρίστες και κυρίως νέους τουρίστες, όπως μας το είπες. Ε, χρειάζεται να ρυθμίσουμε και το ζήτημα της έκδοσης θεωρήσεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, για να αυξήσουμε αυτήν την πελατεία. Ε, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα πρέπει να εξετάσει το συντομότερο δυνατό αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ επίσης, Κάρλο, με τις προτεραιότητες ε, που μα προτείνει σε αυτό το έγγραφο εργασία ε, που υποστηρίζουν και την τουριστική πολιτική των χωρών μας και των περιφερειών μας. Το δικό μας διάβημα έχει κέρια σημασία ώστε να εξασφαλίσουμε ποιότητα, βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και να προωθήσουμε και την εικόνα του τουρισμού στην Γαλλία και σε άλλες χώρες, ε, λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπες, ε, τις κλιματικές αλλαγές ε, που ήδη επηρεάζουν τη συμπεριφορά των τουριστών, κυρίως για τις βραχίες διαμονές σε κάποια άλλη χώρα. Αυτός ο τουρισμός, ο τουρισμός είναι ένας τομέας, ένα προϊόν που δεν μπορούμε να εξάγουμε, γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε, το πολιτιστικό μας κληροδότημα, το, την ε, ποικιλία, την απίστευτη ποικιλία στα ε, ε, τοπία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο φυσικό της περιβάλλον. Θα μιλήσουμε για τον αθλητισμό, για τις μεταφορές, για όλους τους τομείς που ανέφερες εσύ. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε κύριος Δανέλης τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω την, ε, για πρώτη φορά ενασχόληση της Επιτροπής μας με τις ε, επεξεργασίες της Υποεπιτροπής για τον Τουρισμό. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι στην τιτάνια προσπάθεια αναθέρμασης της ανάπτυξης στην Ένωση ο τουρισμός έχει πρωταρχικό ρόλο διότι ξέρουμε ότι παράγει πλούτο και βεβαίως εξασφαλίζει θέσεις εργασίας που άλλες οικονομικές δραστηριότητες δεν μπορούν να κάνουν ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Ε, έτσι η δουλειά της ε, υποεπιτροπής μας για τον τουρισμό νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στην ε, απάντηση και πρακτικών ζητημάτων αλλά και θεμάτων μεθοδολογίας. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες τις οποίες θέτει ο Κάρλο με το έγγραφο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι αποδεκτές δεν θα επαναλάβω αυτά στα οποία αναφέρθηκε και τα οποία θα αποτελέσουν και ζητήματα περαιτέρω επεξεργασίας μας. Ε, νομίζω όμως ότι ο συντονισμός με τις, επιτροπές, τις υπόλοιπες επιτροπές του Κοινοβουλίου αλλά ο συντονισμός επίσης με φορείς και οργανώσεις και οργανισμούς εθνικούς που ασχολούνται με τον τουρισμό θα είναι κάτι το εξαιρετικά χρήσιμο που θα έχει και άμεση ε, αποτελεσματικότητα ε, θα σταματήσω σε δύο ζητήματα τα οποία νομίζω ότι ε, είναι άξια προσοχής μιλώντας για τα μεγάλα θέματα της προσβασιμότητας και της εποχικότητας. Για την προσβασιμότητα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχει η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες ε, τουρισμού βεβαίως, αλλά υπάρχει και το θέμα της προσβασιμότητας και στους τουριστικούς τόπους και κυρίως βέβαια αυτά τα ζητήματα τίθενται στα, όταν μιλάμε για ε, νησιωτικούς τόπους, ε, προορισμούς τουριστικούς ή, ή παρακτίους. Ε, για την εποχικότητα υπάρχει το ζήτημα της προσέγγισης ως φαινομένου οικονομικού αλλά και ως κοινωνικού με την οργάνωση και την δραστηριότητα την κοινωνική. Τέλος, είναι μείζον το ζήτημα της, ε, τελειώνω αυτό, μείζον το ζήτημα της απάντησης στα προβλήματα της ε, της έκδοσης ε, της Visa, ιδιαίτερα για τους προερχόμενους από τις χώρες BRIC. Να μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία εδώ και χρόνια έχει ηλεκτρονική θεώρηση και οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν πολύ εύκολα δεκαετής, ε, πολυετής δηλαδή, θεωρήσεις επισκέψεων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει, όπως έχουμε πει, κατά προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι λαμπρή για την υποπιτροπή μας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με το κείμενο που πρότεινε ο κύριος Φιντάντσα, τον οποίο και ευχαριστώ για το εξαιρετικό του έργο. Εγώ νομίζω πως ε, δεν υπάρχουν στοιχεία να προσθέσουμε εδώ. Γιατί διαφορετικά πρέπει να ξαναγράψουμε την, το, τον φάκελο με στόχο τον ε, τουρισμό. Έχουμε μόλις πέρσι ε, μιλήσει σχετικά. Εγώ νομίζω πως θέλει απλώς ενημέρωση και άρα ως προς αυτό η προσπάθεια της τάσης χώρας αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια αλλά αυτό που θα έκανα θα ήταν να δώσω κάποια μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά την εφαρμογή και, των προθεσμιών. Γιατί εμείς θέλουμε να δεσμεύσουμε τα τρία-τέσσερα χρόνια εργασιών. Από τις παρεμβάσεις όλων δεν κατάλαβα ότι θα πρέπει να είναι πιο σημαντικό αυτό το σημείο στην, στα επιχείρηματά μας. Πέρα από την προσπάθεια που θα κάνει λοιπόν το Προεδρείο ο πρόεδρος Σίμψον και οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών, πιστεύω πως οι πρωταγωνιστές αυτής της Task Force θα πρέπει να παίξουν ακόμα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο να αναλάβουν μια εσωτερική κατανομή των θεμάτων εγώ προτείνω λοιπόν να έχουμε κάποιο περισσότερο χρόνο για να έχουμε στόχο την ετήσια διάσκεψη που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμά μας ως σημείο επαλήθευσης της δουλειάς που έχει γίνει. Ξεκινώντας δηλαδή από το εσωτερικό της Επιτροπής με διάφορα θέματα και φτάνοντας εκείνη τη στιγμή να συνδυάσουμε την κατάσταση πρόοδου που θα είναι το περιεχόμενο αυτού του νέου βήματος που θα πρέπει να εφαρμοστεί στις πολιτικές του τουρισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση, αλλά μερικά πράγματα λείπουν από την έκθεση, διότι μιλήσατε ε, για την αηφορία και τη βιωσιμότητα και το αφήνεται ανοιχτό. Αλλά ξέρουμε ότι ο τουρισμό μπορεί και να καταστρέφει. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στη δικιά σα χώρα και αλλού ε, και θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μα. Γι' αυτό ε, με λυπεί επίσης το γεγονός ότι λείπουν μερικά σημεία. Ας πούμε, έχουμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, ε, πήγα την περασμένη εβδομάδα στην Κροατία σε μια διάσκεψη για τον τουρισμό με τα εμπορικά επιμελητήρια Αυστρίας και Κροατίας και θεώρησαν ότι ορισμένοι πολυδηλατόδρομοι και μονοπάτια θα πρέπει να αυξηθούν, να επεκταθούν το Νοέμβριο βέβαια δεν μπορεί κανείς ε, να κάνει εκεί σκι ε, και είναι χαμηλή περίοδος και πρέπει κάπως να την εκμεταλλευτούν. Είναι θετικό αυτό. Ε, ή έχουμε τους δρόμους της κληρονομιάς, heritage routes, πολιτιστική, φυσική κληρονομιά, ιστορική, βιομηχανική αναδεικνύεται σκεφτείτε τους ιστορικούς σιδηροδρόμους και έτσι δημιουργείται τουρισμός και έτσι αυτό χρειάζεται υποστήριξη. Αυτή είναι βιώσιμη μορφή τουρισμού και λυπάμαι που δεν το γράφετε στην έκθεση. Γενικά για τον οικολογικό τουρισμό, το λέω λέει ο κύριος Φιντάντς αυτό, ε, ε, είναι και αυτό. Ε, για το σήμα, το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι της μόδας τώρα του σειρμού σε πολλές χώρες. Ε, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, το θέμα της θεώρησης διαβατηρίων. Κοιτάξτε μόνο το Καλίνιγκραντ, πόσο δύσκολο είναι να ε, κυκλοφορήσει κανείς και για αυτούς που θέλουν να μπουν και για αυτούς που θέλουν να βγουν από το Καλίνιγκραντ. Το άλλο θέμα, συνθήκες απασχόλησης. Ωραία η φιλικότητα και η καλή συμπεριφορά, μεγάλο ρόλο παίζει και αρχίζει από το αεροδρόμιο, αλλά όταν σου συμπεριφέρονται φιλικά και ευχάριστα ξανάρχεσαι. Ε, για τους πόρους. Από, από την Τεργέστη ε, ε, ξεκινούσε ένα το 1902 που καταργήθηκε το 1930. Είναι πάρα πολύ ωραία η χάραξη. Έχει ε, γέφυρες, ε, κοιλάδες, έχει ε, σύραγγες αλλά δεν μπορεί κανείς να τα επισκεφτεί όλα αυτά γιατί είναι φρικτή υποδομή γύρω-γύρω. Ξέρουμε ότι οι ποδηλάτε, οι τουρίστες με ποδήλατο ε, ημερησίως δαπανούν περισσότερα χρήματα από εκείνου που είναι με αυτοκίνητο. Ευχαριστώ, Μάικλ. Είσαι βέβαιος ε, από εκείνοι που, επισκέπτονται ε, τους σιδηροδρόμου, τους ιστορικούς, δεν είμαι βέβαιο. Ο κύριο Πίρκερ, ο κύριος Φιντάνσα έκανε ένα πολυετές πρόγραμμα νομίζω μας παρουσίασε μόλις με πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά σημεία μόνο. Αυτό με την ετήσια διάσκεψη έχει νόημα, μεν, αλλά μάλλον στην αρχή και όχι στο τέλος του έτους, όπως είπε ο κύριος Ουτζίας. Δηλαδή, ε, να μην έχουμε επικαλύψεις και διπλή δουλειά με συγκεκριμένους στόχους. Και η επιτυχία τέτοιων διασκέψεων και συνεδριών εξαρτάται από την σύστασή τους και από τα μέλη τους. Ας πούμε, επιχειρηματίες που έχουν υποδειγματική δραστηριότητα, ας πούμε τουρισμός για ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα ή εμπειρογνώμονες. Ε, πολλές φορές είναι μεγάλες οι προσδοκίες, αλλά θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό και το αποτέλεσμα τέτοιων διασκέψεων. Ένα δεύτερο που θέλω να αναφέρω τονίζεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να τονωθεί, λέει. Ε, ε, χρειαζόμαστε ε, να αναλύσουμε τις διάφορες τάσεις, όπως έχει να κάνει η φύση με την σωματική δραστηριότητα, και στο νότο της Ευρώπης ε, μπορούμε να προωθήσουμε άλλες μορφές. Επίσης στην ε, ανταγωνιστικότητα ανήκει και μια ποιοτική, καλύτερη προσφορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προτείνει και ο κύριος Φιντάντσα και νομίζω ότι θα πρέπει να το ε, αξιοποιήσουμε. Κάτι άλλο που ανήκει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι και το διαδίκτυο και ε, τα εισιτήρια, ε, ένα ενιαίο εισιτήριο ε, που μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς, σύνδεση δηλαδή αεροπορικών με σιδηροδρομικά εισιτήρια λεωφορείων και τα συστήματα ταξινόμησης επιτέλους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν θέλουμε να έχουμε μία μάρκα, ένα σήμα Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχει και συγκρισιμότητα εσωτερική για δηλαδή το σύστημα των αστέρων, των ξενοδοχείων κτλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Κάρλο είναι ιδιαίτερα μετριοπαθή όταν παρουσιάζει το έγγραφό του ω έγγραφο εργασία. Έχει τόσο πολύ υλικό που ουσιαστικά πρόκειται για πλήρε έγγραφο χάραξη πολιτική. Ε, ε, είναι φάνταστο αλλά και πρακτικό ταυτόχρονα, πλούσιο και μα προσφέρει πολλά. Λοιπόν, ε, για να αποφύγουμε επικάλυψη, δίκιο έχει ο Κάρλο ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε τι κάνουν και εκείνοι, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί και πώ μπορούμε να αλληλοσυμπληρωθούμε. Ε, για την Κυπριακή Προεδρία τώρα. Η Κύπρος όπως και η Ιρλανδία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, οπότε το ζήτημα είναι σημαντικό και για αυτούς. Ε, και ο τουρισμός και η γεωργία είναι δύο τομείς που έχουν πληγεί σημαντικά και στις δύο οικονομίες. Εμείς τι κάνουμε στην Ιρλανδία. Ε, πάνω από 40 ε, εκατομμύρια Ιρλανδοί διαβιούν στη ΣΥΠΑ και το 2013 έχει αναδειχθεί στο έτος της συγκέντρωσης, της συναισθίασης. Από όπου και αν έρχονται, είπα Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Αυστραλία, όλοι οι Ιρλανδοί ομογενεί να επιστρέψουν επιστρέψουν από το αρχικό σημείο της μετανάστευσης. Σε σχέση με αυτά που μας είπε ο Μάικλ κρεαμέρε για το, τους πολιτιστικούς δρόμους ε, και τα λοιπά. Ε, στο 3β Βλέπουμε μία απάντηση, διότι για να διαφυλάξουμε, λέει στο σημείο 3, την ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να προωθήσουμε τον επιστημονικό τουρισμό, τον ποδηλατικό τουρισμό, θαλάσσιο τουρισμό, παράκτιο τουρισμό, ε, τουρισμό της υπαίθρου κτλ. Ε, υπάρχουν όλα αυτά, μα έκλειδεσμε. Ε, και πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό το έργο μας, διότι είναι εξαιρετικά πλούσιο αυτό το έγγραφο. Ευχαριστούμε, κυρία Εστέρας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Κάρλο Φιντάνσα. Είναι πάρα πολύ καλό το έγγραφό του και πάρα πολύ καλά δομημένο. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω τα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, για το συντονισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τον εγκάρσιο χαρακτήρα, τον οριζόντιο του τομέα. Ό,τι και αν αποφασιστεί, ε, σε οποιαδήποτε επιτροπή του Κοινοβουλίου αφορά τον τουρισμό, ε, το φαγητό, το ποτό, η φόρη, η υγεία, οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, τα νοσοκομεία, τα πάντα, η εκπαίδευση, με κάποιο τρόπο αφορούν τον τουρισμό. Γι' αυτό, ε, αυτό τον καιρό συζητείται ένα θέμα που είναι ο θόρυβος ή το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας που επηρεάζει πάρα πολύ τον τουρισμό. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ότι είναι οριζόντιος χαρακτήρας να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Όποια απόφαση ε, και αν πάρουμε ή οποιαδήποτε απόφαση που παίρνουμε στις επιτροπές μας αφορά την ποιότητα του τουρισμού, σε ό,τι αφορά τον εποχιακό χαρακτήρα. Αυτό συνδέεται κυρίως με τη διαφοροποίηση. Δηλαδή, πολύ ωραία λέγει το έγγραφο ότι ο εποχιακός χαρακτήρας μπορεί να διέπεται από διάφορα στοιχεία. Αλλά όταν έχεις ένα τουριστικό προορισμό που είναι θάλασσα και ήλιος, ε, πρέπει να δεις πώς μπορείς να το διαφοροποιήσεις και να προσφέρεις και άλλα πράγματα. Ε, τουριστικές διαδρομές, όπως είπε και ο κύριος Κράμερ, ε, για τον ποδηλατικό τουρισμό, το συνεδριακό τουρισμό, τον υγειονομικό, τον πολιτιστικό, της πολιτιστικής κληρονομιάς, όλα αυτά νομίζω πρέπει να μπουν σε δύο εκθέσεις. Το ένα να είναι τουρισμός και προσβασιμότητα και το άλλο ε, τουρισμός και διαφοροποίηση και εποχικότητα. Γιατί αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε ένα διαχρονικό τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όπου είναι μικρή η σεζόν, κλείνουν τα ξενοδοχεία, ε, κλείνει η υπόλοιπη υποδομή, οπότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση τώρα. 80 εκατομμύρια είναι οι Ευρωπαίοι με προβλήματα αναπηρίας. Είναι σημαντική ομάδα του πληθυσμού και ε, φέτος έχουμε βαφτίσει και το έτος αυτό, έτος της ενεργούς γύρασης και ηλικιωμένοι είναι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού Και τα ξέρει αυτά και ο κύριος Φιδάντσα. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να τυποποιήσουμε τα σήματα, ε, τα σύμβολα ε, για να ξέρει κάποιος αν είναι προσβάσιμο ένα ξενοδοχείο ας πούμε ε, για άτομα με αναπηρία. Ούτε καν τα σύμβολα δεν είναι ενιαία για να μπορέσουμε να τα ερμηνεύσουμε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι στον κύριο Φιδάνσα. Ο κύριος Κομουτσάκος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην προηγούμενη και πρώτη συζήτησή μας ε, όταν ε, συστήσαμε, όταν συστήθηκε η Task Force για τον τουρισμό είχα την ευκαιρία να πω ότι θα ήταν καλό να υπάρξει ένας οδικός χάρτης, ένας οδικός άξονας, ένας οδικός χάρτης με ορισμένες συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες και επομένως δεν μπορώ παρά να καλωσορίσω, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ε, τον ε, αγαπητό συνάδελφο κύριο Φιντάντζα για την πρόταση που ε, καταθέτει, για τις σκέψεις που σήμερα καταθέτει. Ε, ακολουθούν ακριβώς αυτή τη λογική της κατανομής μέσα στον χρόνο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για να ενισχύσουμε την εργασία που πρέπει να κάνει η Task Force για τον τουρισμό είναι η σωστή προσέγγιση, έχει την απόλυτη υποστήριξή μου και χαίρομαι γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η στήριξη δίδεται και από το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων ε, και αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουμε. Δύο μόνο θέματα πολύ επιγραμματικά. Η εποχικότητα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, πρέπει, είναι πολύ δύσκολο να περάσεις ε, την τουριστική βιομηχανία και τη φιλοσοφία του τουρισμού από την παραδοσιακή ροή σε συγκεκριμένους χρόνους και περιόδους της, ε, του έτους σε ολόκληρο το έτος και νομίζω ότι είναι ένα τομέας στον οποίο πρέπει ειδικά να επικεντρώσουμε την προσοχή μας διότι απαιτεί αλλαγή και νοτροπίας και υποδομών και management είναι μεγάλη, ενώ εύκολα λέγεται, ε, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Το δεύτερο σημείο, και ε, θα σταματήσω με αυτό, είναι η πρόταση για, την ετήσια, για το ετήσιο συνέδριο για τον τουρισμό, το Annual Conference. Εδώ θα συμφωνήσω απολύτως με την παρατήρηση του συναδέλφου κύριου Πίρκερ, ότι αυτή η ετήσια σύνοδος, αυτό το ετήσιο συνέδριο για τον τουρισμό, πρέπει να γίνεται στην αρχή του χρόνου, στην αρχή του τουριστικού έτους. Ο Μάιος είναι αρκετά κοντά στις παραδοσιακές περιόδους τουρισμού και πάντως έχουν περάσει πέντε μήνες. Ε, πέντε μήνες από την έναρξη του χρόνου. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνάδελφο κύριο Φιντάντζα να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή η πρώτη ετήσια σύνοδος να γίνει όχι αργότερα από το τέλος Φεβρουαρίου ή μέσα Μαρτίου σε απότατο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. For myself, I'll θέλω να σχολιάσω το θέμα της διάσκεψης, επιτρέψτε μου, γιατί λένε όλοι ότι είναι μια υπέροχη ιδέα, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος που θα βρούμε τα λεφτά ή πώς ε, θα προσφέρουμε τα απαραίτητα για τη διάσκεψη. Ίσως, ε, Κάρλος, θα μπορούσες ε, να το επανεξετάσεις αυτό το θέμα, να μιλήσεις για σεμινάριο, για ανταλλαγή ιδεών, brainstorm, τέλο πάντων, οτιδήποτε. Πάντως, αυτό δεν εντάσσεται στην εντολή της Επιτροπής μας. Δεν μπορούμε να διοργανώσουμε εμείς κάτι τέτοιο, ούτε από οικονομικής πλευράς, ούτε από πλευράς προσωπικού, αλλά ούτως ή άλλως θα επανόλθουμε σε αυτό το θέμα για τα υπόλοιπα τώρα σημεία. Είναι εξαιρετικά εξαιρετική ποιότητα το έγγραφο. Είναι ένα σημείο κίνησης ένας οδικό χάρτης σε πού είμαστε τώρα, πού πάμε κτλ. Ο Μάικλ δίκαια προβάλλει ενστάσει. Τα ίδια είπα και εγώ για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ε, αν δεχθούμε ότι ο ποδηλατικό τουρισμό, ε, το βιομηχανικό κληροδότημα έχουν σημασία, ε, λοιπόν πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και να αναπτύξουμε ευρωπαϊκά δίκτυα, να χτίσουμε κάτι γύρω από αυτές τις ιδέες. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για παράληψη. μέσα στο έγγραφο αυτό απαριθμούμε απλώς ε, τα μελλοντικά μας βήματα. Είναι εξαιρετικό το έγγραφο και θα πρέπει να το δείτε ως ε, οδηγό. Δεν είναι <laughs> οι δέκα εντολές. Ε, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε την πολιτική τουρισμού σε συνεργασία με τις συναρμόδιες γενικές και σε διευθύνσεις ε, και καλό θα ήταν να το δούμε μέχρι το τέλος του έτους και όχι στις αρχές του επομένου. Πρέπει να θέσουμε σε κίνηση το μηχανισμό γιατί είναι άνευ προηγουμένου. Πρώτη φορά ασχολούμαστε με τέτοιο ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είχαμε αρμοδιότητα καν μέχρι τη συνθήκη της Λισαβόνας για τα θέματα τουρισμού και ε, σε αυτό έγκυται και ένα από τα προβλήματα όταν μιλάμε για την ταξινόμηση των ξενοδοχείων. Το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να εκχωρήσουν τις αρμοδιότητές τους και έκαναν ό,τι έκριναν σωστό. Τώρα όμως πρόκειται για νέο στοιχείο. Ξαναλέω, τώρα έχουμε πλέον αρμοδιότητα και Επιτροπή πως ε, τα Γιάννη και οι υπόλοιποι προωθούν το ζήτημα και ε, καλά θα κάναμε στο Κοινοβούλιο ε, να ακολουθήσουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το έγγραφο ως βάση. Δεν είναι θέσφατα αυτά που λέει, το ξαναλέω, δεν είναι δέκα εντολές. Θα είναι μια βάση για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Σας ευχαριστούμε πάντως και Φιντάνση και ευχαριστούμε και το προσωπικό που συνέβαλε στην κατάρτιση του εγγράφου. Κύριε Ζώτνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να να πάρει το λόγο τώρα. Πάντοτε είσαστε πάρα πολύ σύντομο και λακωνικό. Ελπίζω να επαναληφθεί και σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλου. Χαίρομαι ιδιαίτερω που με καλέσατε για να σχολιάσω αυτό το σημείο τη διάταξη. Είναι επίκαιρο το ζήτημα, διότι καλό θα ήταν να γνωρίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την έγκριση τη ανακοίνωση τον Ιούνιο εφαρμόζουμε και τι 21 και πλέον δράσει που κατονομάζονται μέσα στην ανακοίνωση ανακοίνωση είναι σε διαδικασία εφαρμογή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και ένα ολόκληρο φάσμα επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δεν μιλάμε μόνο για αυτέ τι δράσει, αλλά και για νέε δράσει που ανέκυψαν του τελευταίους μήνε και χρόνια που αποτυπώνονται σε έναν χάρτη ε, που ε, δημοσιεύουμε τακτικά στην ιστοσελίδα μας. τελευταία δημοσίευση έγινε το Μάιο και την την επόμενη εβδομάδα θα επικαιροποιήσουμε ε, την ιστοσελίδα προετοιμαζώντα ε, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Τουρισμό, ετήσια δηλαδή συνεδρίαση, όπου όλοι οι φορεί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα του τουρισμού θα συνεδριάσουν σε τρει εβδομάδε στην Κύπρο. Οι βασικές μας δράσεις ε, σχετίζονται με τρεις βασικά τομείς. Πρώτον, αύξηση της ζήτησης για τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ιστορικό των κρατών μελών και κυρίως ε, στις ε, χαμηλές περιόδους. Θέλουμε να διευρύνουμε την υψηλή περίοδο ή να μειώσουμε την χαμηλή και στη συνέχεια να αυξήσουμε τις ροές τουριστών από τρίτες χώρες καθώς και να ασχοληθούμε με τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Η δεύτερη δράση η διαφοροποίηση της προσφοράς και αναβάθμιση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα και σε επίπεδο ιδιώτη και σε επίπεδο επιχειρήσεων και έτσι εν συντομία μπορώ να σας αναφέρω τις βασικές πρωτοβουλίες για αυτό το ζήτημα, για ε, το, το IEC, το πρόγραμμα προσβασιμότητας και ούτω καθεξής. Στην ε, συνέχεια ε, προσπαθούμε στον τομέα του τουρισμού, όπως είπατε και εσείς, να αντιμετωπίσουμε το θέμα εργασίως. Ε, δηλαδή, ο τουρισμός θέλουμε να ενταχθεί και στις πλέον σημαντικές πολιτικές για τις θεωρήσεις, για τις μεταφορές, για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό, για την εσωτερική αγορά και ούτω κάθε εξής. Και στη συνέχεια, σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαθέτουμε, συγκεκριμένα να έχουμε ένα συγκεκριμένο μικρό ταμείο για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και τα μέσα που ανέφερε ο Κάλλος Φιντάνσε για τη χρηματοδότηση, αλλά ε, ε, είτε μιλάμε για τα διορθωτικά ταμεία, είτε για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, για το Ταμείο Αλίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και τέτοιες πηγές χρηματοδότησης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, προσπαθώ όμως παρόλα αυτά να ανατρέξω όλα τα σημεία και να σας ενημερώσω για κάθε ένα από αυτά τι έχουμε κάνει, αυτά τα σημεία δηλαδή που παρουσίασε ο Κάρλος Φιντάνσα στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων ε, για αυτή την πολιτική προώθηση της συνεργασίας. Καλούμε <clears throat> το Κοινοβούλιο σε όλες τις ε, εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και φυσικά θέλουμε να μετάσχουμε σε αυτή την ετήσια διάσκεψη, συνεδρίαση όπως την πείτε, ό,τι και αν διοργανώσετε, καλό θα ήταν να μας καλέσετε για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις, για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ε, δεύτερον, τουρισμός για όλους προσβασιμότητα. Ε, μέσα στην πρωτοβουλία μιλάτε για προπαρασκευαστική δράση που όμως ήδη υλοποιείται, έχει δρομολογηθεί και έχουμε ένα εκατομμύριο για το 2012 ε, και ε, προτάθηκε παράταση και για το 2013 ε, με διάφορες πρωτοβουλίες ώστε να προσδιορίσουμε ποια είναι ποιες είναι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες προσφοράς και ζήτηση για να βελτιώσουμε την πρόσβαση ε, στα τουριστικά αξιοθέτα και τους τουριστικούς προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώνουμε και ένα βραβείο για, τις, ε, για να επιβραβεύουμε οργανώσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Στη συνέχεια ολοκληρώσαμε την προσκευαστική δράση Καλύψω ε, το πρώτο στάδιο και παρατή δίνουμε τώρα αυτή την πρωτοβουλία σε, με μεγάλη δυσκολία σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αυτέ οι πρωτοβουλίε ε, με σημείωσαν αρκετή επιτυχία και ο Επίτροπο ε, Ταγιάννη τώρα ε, πρότεινε μια νέα δράση για του ηλικιωμένου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να ε, προωθήσουμε το, ανταλλαγέ ανταλλαγές ηλικιωμένων στη χαμηλή τουριστική περίοδο, αυτά για την εποχικότητα Έγινε μια συνεδρία είναι από δύο εβδομάδε ε, και η Ευρωπαϊκή Μέρα τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου ε, ήταν άλλη μια ευκαιρία για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Στη συνέχεια, διαφοροποίηση και βιωσιμότητα. Φυσικά, μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Καλύψε και σε προηγουμένων ετών σε σχέση με την ε, προπαρασκευαστική δράση για την βιωσιμότητα, για τους ποδηλατοδρόμους, το ποδηλατικό τουρισμό και δύο διαγωνισμούς ε, ξεκινήσαμε. Το δεύτερο ε, τώρα ξεκίνησε για το 2012. 58 προτάσεις λάβαμε για τα βιώσιμα τουριστικά προϊόντα στον τομέα του αθλητισμού, περιπετειώδους τουρισμού, ποδηλατικού τουρισμού κτλ κτλ. Θα θυμάστε επίσης ε, ότι μας είχατε δώσει και μια άλλη γραμμή του προϋπολογισμού, μια άλλη προπαρασκευαστική δράση για την προώθηση ε, της, ε, του βιομηχανικού κληροδοτήματος και του τουρισμού. Έκλεισε ένας διαγωνισμό διαγωνισμός την περασμένη εβδομάδα και λάβαμε 50 προτάσεις, οπότε μην ανησυχείτε, ασχολούμαστε με αυτό το στοιχείο της διαφοροποίησης της προσφοράς και θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε στις αρχές του 2013 για αυτά. Τέταρτος βασικός τομέας, ε, ε, δηλαδή η προσέλκυση ροών από τρίτες χώρες και συγκεκριμένα πολιτική θεωρήσεων. Θα γνωρίζετε ότι ε, συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και με την κυρία Μάλστρομ και τον κύριο Ταζάνη και τις επόμενες ημέρες, ή τέλος πάντων κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, θα εκδώσουμε κοινή ανακοίνωση μετά από έγκριση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα ενέχει διάφορες οποια θα ενεχει διάφορε βελτιωσεις και απλούς ε, του κώδικα θεωρήσεων υπάρχουν ακόμη δυνατότητες ε, με τον τωρινό κώδικα ε, να απελευθερώσουμε το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων μειώνοντας προθεσμίες για να κλείσει κάποιος ραντεβού ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε όλα τα έντυπα σε όλες τις απαιτούμενες γλώσσες. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα δείτε στην ανακοίνωση επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΧΟΜΑ, θα συμμετάσχουμε στην επερχόμενη αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων που θα λάβει η χώρα το 2013 και ήδη έχουμε αρχίσει τα προπαρασκευαστικά στάδια των μελετών για να προετοιμάσουμε την αναθεώρηση του κώδικα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν υπάρχουν στρατηγικές για την αγορά. Ξέρετε ότι δρομολογήσαμε εκστρατεία ενημερωτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις τέσσερις μεγάλες αγορές, μεταξύ των οποίων Χιλή και Αργεντινή. Έχουμε προπαρασκευαστική δράση και επιδότηση προς την ITC, την οργάνωση που ε, εκπροσωπεί όλους τους οργανισμούς τουρισμού που θα αναλάβει την αποκοινού προώθηση του τουρισμού με συμμετοχή των εθνικών φορέων αλλά και σε συνεργασία με τρίτες χώρε Καναδάς, τα κτλ. Επενδύσεις για την ποιότητα τέλος, ε, ε, εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας ε, και στο ε, είμαστε στο τέλος ε, της εσωτερικής διαδικασίας προετοιμασίας για ένα συνολικό σύστημα, μια συνολική πρωτοβουλία για τα ποιοτικά σχέδια που υπάρχουν ή που θα αναπτυχθούν είτε σε εθνικό είτε σε κλαδικό επίπεδο, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα γενικό σήμα ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιολόγηση αντικτύπου μελετή έχει κατατεθεί ήδη στο Συμβούλιο και το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το τέλος τέλος 2012 θα έχει εγκρίνει ε, την πρόταση για το σήμα και ελπίζω στις αρχές του 2013 να φτάσει στο Κοινοβούλιο. Για τους πόρους και θα κλείσω με αυτό, Έχουμε στην, ε, ε, την πρότασή μας, τώρα το μπαλάκι όμως είναι στο γήπεδο του ε, Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το κόσμο. Έχουμε κάνει προτάσεις για το τουρισμό, ξέρετε, το γνωρίζετε πολύ καλά και συζητούνται εδώ στο Κοινοβούλιο κάποιες σχετικέ συμβαστικές τροπολογίες. Δεν θα είναι εύκολες συζητήσεις με το Συμβούλιο, διότι κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν να αφαιρθεί ο τουρισμός στην πρόταση κόσμο. αλλά το σημαντικό είναι να προβάλλουμε τον τουρισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά μέσα. Στην πρόταση τη Επιτροπή καταφέραμε να αναφέρουμε τον τουρισμό στο Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, στο Ταμείο Ανάπτυξη Πέθρου, στο Γεωργικό Ταμείο, σε όλα τα πολιτικά προγράμματα, καθώ και στο πρόγραμμα εξωτερική δράση Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη υποστήριξη από πλευρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα τα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι ευπρόσδεκτη και είμαστε στη διάθεσή σα αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσει ή αν θέλετε να διοργανώσετε κάποια συνεδρία, ώστε να υψέλθουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε σα υπενθυμίζω όμως ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίε ε, τακτικά ε, αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας ε, και είναι διαθέσιμες και για εσά και για όλους μας και κυρίως για του εμπλεκόμενου φορείς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κάρλο, έχουμε καθυστερήσει τώρα. Εγώ προτείνω το εξή να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται από την Επιτροπή το έγγραφό σου και να βασιστούμε σε αυτό για να προχωρήσουμε. Θα ελέγξουμε αυτό το θέμα της διάσκεψης, γιατί ξέρω ότι είναι πηγή ανησυχιών. Θέλεις να προσθέσεις κάτι εντάχει, σε παρακαλώ. Ναι, σύντομα να πω κάτι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τα καλά τους λόγια. Με χαροποιεί ότι όπως υπογράμμισαν ε, όλοι θέλουν να συνεργαστούν ε, και μάλιστα να προβλέψουμε και μια κατανομή των θεμάτων γιατί είναι πολύ σκόπιμα πέρα από τη δουλειά που εγώ μπορώ να κάνω και που ευχαρίστως το κάνω και που μια που το εκτιμάτε και όλα ακόμη περισσότερο με χαροποιεί αυτό αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μέσω της ενεργής συμμετοχή, ενεργού συμμετοχής όλων σας για το θέμα της ε, συνάντησης με την Κυπριακή Προεδρία που υπογράμμισε και ο συνάδελφος Χίγκινς θα το προσπαθήσω δυστυχώς όταν ξεκινήσαμε το εξάμεινο της Προεδρίας, περίμενα να δοθεί κάποια έμφαση στις πολιτικές τουρισμού. Αντιθέτως δεν το είδαμε αυτό. Όταν ακούσαμε δηλαδή τον Υπουργό Τουρισμού, δεν ξέρω, ίσως ήταν λίγο αργά. Και όσον αφορά την ετήσια διάσκεψη, θα το επαληθεύσουμε όσον αφορά τα οργανωτικά ζητήματα με τον Πρόεδρο. Εγώ είμαι υπέρ να γίνει λίγο πριν από την αρχή της σεζόν να κάνουμε και σημαντικές εντωμεταξύ ενημερώσεις. Θα πρέπει να προβλέψουμε κάποια συγκεκριμένη στιγμή για την ενημέρωση για τις 21 δράσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε κάποια θέματα και να τελειώσω, Πρόεδρε, ζητώντας σας την εντολή για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το θέμα των τροπολογιών για το κόσμο, για να μπορέσουμε να στείλουμε και μια επιστολή στο όνομα της Task Force, υποστηρίζοντας την θέση που ήδη είχαμε στην έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τη γραμμή χρηματοδότηση του τουρισμού, επαναλαμβάνοντας δηλαδή στους συναδέλφους της Επιτροπής Ήτρη τη σημασία αυτή στις αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν, θα ήθελα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες, αφού θα προχωρά σιγά σιγά και η διαπραγμάτευση για τις τροπολογίε. τροπολογίες. Να μπορέσω να διατηρήσω αυτή τη θέση, όπως κάναμε μέχρι στιγμής, στο όνομα όλων. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα. Να σας δώσουμε αυτή την εντολή σε σχέση με την επαφή με τις υπόλοιπες επιτροπές. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η πρώτη ανάγνωση για το θέμα του ελέγχου των πλοίων από το κράτος Λιμένα. Εγώ είμαι ο εισηγητής. Θα ήθελα να σας πω τα εξής σε σχέση με το τι περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο εξής. Καταρχήν έχουμε την σύμβαση της θαλάσσης για τους ναυτικούς ε, που υιοθετήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας το 2006. Οι συνθήκες απασχόλησης κατάλυσης, ε, αναψυχής, ε, ιατρικής περίθαψης κτλ. κτλ. αναφερόταν εκεί. Ήταν η πρώτη συνολική σύμβαση ναυτικής ε, εργασίας που καλύπτει 1,2 εκατομμύρια ναυτικούς παγκοσμίω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας για 30 φορά κύρωσε την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας φέτος στις 20 Αυγούστου ώστε αυτή να αρχίσει να ισχύει στις 20 Αυγούστου 2013. Πολλά κράτη, όπως η Κύπρος, Δανία, Λετωνία, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία, ήταν μεταξύ των πρώτων 30 χωρών που προσχώρησαν σε αυτήν, όπως και η Κροατία, η Νορβηγία και η Ελβετία. Αυτό που με εντυπωσιάζει για όλα αυτά είναι ότι ενώ υπάρχουν ε, χώρες χωρίς ε, θαλάσσια σύνορα όπως το Λουξεμβούργο και η Ελβετία που συνυπογράφουν αυτή τη σύμβαση οι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τη συνυπογράφουν. Η ευρωπαϊκή τώρα νομοθεσία ήδη έχει ευθυγραμμιστεί με τις περισσότερες ε, σχετικές διατάξεις της ε, Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας μετά από συμφωνία ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους. Ωστόσο, δεν είχαν την εξουσία, την αρμοδιότητα να συμπεριλάβουν τις διατάξεις επιβολής που συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο 5 της ε, Σύμβασης. Οπότε, η, πρόταση με την οποία ασχολούμαστε τώρα απαιτεί αυτή την επιβολή και αφορεί αφορά την ευθύνη του κράτους σημαία που απορρέει από αυτήν. Θέλουμε να καθιερωθούν ελάχιστα πρότυπα για τι συνθήκε εργασία και διαβίωση επιτοπλίων. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα τη ναυτιλία, τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ισχύουν για όλο τον κλάδο. Τα πλοία που δεν πληρούν τα σχετικά πρότυπα είναι μη αποδοκτά όσο, τόσο σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων, όσο και σε σχέση με την ασφάλεια, την προστασία από παράνομε ενέργειε και την προστασία του περιβάλλοντο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, να προσφέρει του μηχανισμού ώστε να, να εξασφαλίζεται ότι τα πλοία συμμορφώνονται με του σχετικού κανόνε, άσχετα με την εθνικότητα των ναυτικών και την, το κράτος σημαίας του πλοίου. Επιπλέον θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μην υποβαθμίζονται οι συνθήκες εργασίας εις ε, βάρος των πληκτικών που προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες όπως προβλέπονται από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Τα δε πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους σημαίας που δεν έχει, κυρω, έχουν, έχει κυρώσει τη δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα από τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους που την έχουν κυρώσει. Το Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει τονίσει τη σημασία ενίσχυσης της ελγιστικότητας των ναυτικών επαγγελμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί των πλοίων. Βέβαια είναι ευπρόσδεκτε οι ελάχιστε διεθνεί προδιαγραφέ, ωστόσο θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην αποτελούνται αυτά ω ε, ε, δικαιολογία για να υπονομεύσουν τα υφιστάμενα επίπεδα προστασία που παρέχονται βάσει τη Ευρωπαϊκή Κοινωνική Νομοθεσία. Εκτό από τι τροπολογίε που καθιστούν σαφέ ότι τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα δεν δικαιολογούν την υπανόμευση των υπαρχών των ευρωπαϊκών προτύπων, όταν τα πρότυπα αυτά είναι υψηλότερα, ορισμένε άλλε τροπολογίε επιδιώκουν την περαιτέρω ευθυγράμμιση τη οδηγία για τον έλεγχο από το κράτο λιμένα με το κείμενο τη Σύμβαση Ναυτικών Εργασιών. Επίσης, ε, μια σειρά τροπολογιών επιδιώκει να διασφαλίσει ότι πληροφορίε θα διαβιβάζονται στη Διεθνή Οργανισμό εργασία και άλλες ε, για να ενισχύσουν τις ζήτησεις που αφορούν το απόρριτο καταγγελιών. ώστε οι ναυτικοί να μην διστάζουν να υποβάλουν καταγγελίες λόγω των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών ή ακόμα και λόγω ύπαρξης μαύρου, μαύρης λίστας. Τα κράτη-μέλη είχαν από το 2006 για να προετοιμάσουν την απαραίτητη εθνική νομοθεσία και η περίοδος μεταφοράς θα πρέπει να σμεκρινθεί ώστε τα κράτη να έχουν συμμορφωθεί πλήρως όταν θα αρχίσει να ισχύει τον Αύγουστο του επόμενου χρόνου η Σύμβαση ναυτικών, ε, ε Ναυτικής Εργασίας. Η Οδηγία 2009-16 τροποποιείται για πρώτη φορά μετά την έναξη τη Λισαβόνα και απαιτούνται νέοι κανόνε για την έκδοση κατεξοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Ω προ αυτό ε, το σημείο έχουμε τη συνήθη θέση του, του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η εξοδότηση δεν πρέπει να παρέχεται επαόριστο ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τι εξουσίε τη πριν ανανεωθεί η εξουσιοδότησή τη. Παρόλο που είναι σημαντική η έγκαιρη κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, ε, δεν, είναι, δεν αρκεί. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προσλάβουν επαρκή αριθμό επιθεωρητών με κατάλληλε δεξιότητε, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αξιολογούν τι ειδικέ εργασίες και διαβίωση των ναυτικών ε, στα πλοία. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατάρτιση των επιθεωρητών και στο συντονισμό αυτών, ώστε να διεξάγουν ε, του ελέγχου τη Σύμβαση Ναυτική Εργασία. Ε, υπ' αυτή την ε, νέα σα υποβάλλω αυτή την έκθεση και κύριε Κουμουτσάκο έχετε εσεί πρώτο τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα, είμαι, είμαι σύντομος και ελπίζω ουσιαστικός να ξεκινήσω λέγοντας ότι ορθώς προχωράμε σε τροποποίηση της οδηγίας του 2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος Λιμπενά. Ε, αυτό έγινε επιτακτικό μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, της MLC, από περισσότερα από 30 κράτη και επομένως η Σύμβαση πλέον μπορεί να τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον προσεχή Αύγουστο του 2013 δηλαδή. Επομένως είναι επιτακτικό για την Ένωση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει στην τροποποίηση της οδηγίας του 2009. Ε, η τροποποίηση βέβαια αυτή επικεντρώνεται στον ειδικό τέταρτο τίτλο της σύμβασης, της MLC, εκείνον δηλαδή που αφορά την εφαρμογή και συμμόρφωση με τα όσα προβλέπει το, το υπόλοιπο κομμάτι, τα άλλα τέσσερα τμήματα της σύμβασης αυτής. Όπως ε, κύριε Πρόεδρε και όσοι συγητής αναφέρετε στην αιτιολογική σας έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα ένθερμος υποστηρικτής της θεσμοθέτησης μέτρων για την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων επιτομπλίων. Επομένως, αυτή η σταθερή μας θέση πρέπει να είναι και καθοδηγητική για την δουλειά που πρόκειται να κάνουμε στην διαδικασία της τροποποίησης της οδηγίας. Άλλωστε, ε, αυτή ήταν η θέση του Κοινοβουλίου γιατί πιστεύουμε ότι η υποστήριξη μέτρων ελαχίστων προτύπων για τις συνθήκες εργασίας και τις διαβίωσης των ε, επιτομπλίων πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην επίτευξη ενός άλλου στρατηγικού μας στόχου που είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας του ναυτικού επαγγέλματος για τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επιτοπλίων. Επομένως, ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω ότι συμφωνώ με τη γενική κατεύθυνση των, ε, όσων μας παρουσιάζεται σήμερα. Ε, θα πρέπει όμως να επισημάνω και δύο ε, γενικές παρατηρήσεις ότι στις τροπολογίες μας πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το βάρος ε, της, ε, του ελέγχου συμμόρφωσης θα πρέπει πρωτίστως να το έχει η εταιρεία και το κράτος σημαίας. Εκείνοι έχουν τη μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης. Το κράτος λιμένα έχει μια αρμοδιότητα συμπληρωματική ελέγχου. Αυτό όμως δεν την κάνει και λιγότερο σημαντική αλλά πάντως στην ουσία της παραμένει συμπληρωματική. Την κύρια ευθύνη έχουν τα κράτη σημαίας και εταιρείε. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο ε, ζητήματα, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ότι εάν επιβαρύνουμε, εάν ζητάμε από τους επιθεωρητές επιπλέον γνώση και κατανόηση των θεμάτων, αυτό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα και μιας εκπαίδευσής τους διότι γίνεται πιο σύνθετη η αποστολή τους. Και εδώ καλό είναι να συγκρατήσει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα η ΕΜΣΑ να καλύψει αυτή την ανάγκη και εν πάση περιπτώσει να αναζητήσουμε ένα ρόλο της προς αυτή την κατεύθυνση διότι το έργο των επιθεωρητών γίνεται εξαιρετικά απαιτητικό. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι το άλλο σημείο, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να υπερβούμε την λογική της παρακολούθησης των ελαχίστων, ε, του ελαχίστου κοινού παρονομαστή. Κοιτάξτε, αν οι επιθεωρήσεις γίνουν υπέρ των δέων λεπτομερείς, έχουμε δύο πιθανά προβλήματα. Πρώτον, να μην είναι τελικά ουσιαστική η επιθεώρηση, να χάνεται πολύτιμος χρόνος ακόμα και να οθήσουμε σε μια συμφόρηση των λιμένων καθώς οι επιθεωρήσεις θα κρατάνε πάρα πολύ. Επομένως πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής παρακολούθησης της εφαρμογής των όσων προβλέπονται στην MLC αλλά και ταυτόχρονα μιας ευελιξίας που θα διασφαλίζει δύο πράγματα. Και τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων στα πλοία, αλλά και δεν θα επιτρέπει μία παράλογη, αν θέλετε, επιβάρυνση αυτής της διαδικασίας. Με αρνητικά, πιστεύω, αποτελέσματα ε, στην, ε, στην όλη διαδικασία. Με αυτές τις βασικές σκέψεις, ε, κύριε Πρόεδρε, προτίθεμαι να καταθέσω ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες πιστεύω ότι ε, θα κάνουν το ήδη πολύ καλό δικό σας κείμενο ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ταυτόχρονα τον Πρόεδρό μας για την έκθεσή του. Πάντα λέω ότι μ' αρέσουν οι εκθέσεις του κυρίου Σίμψον. Εχθές γύρισα από την Κύπρο Είχαμε μια διημερίδα για τη λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη και την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τη μεταξέλιξή της και συμφωνούμε όλοι ότι τα θαλάσσια επαγγέλματα τα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο γιατί θα αυξηθεί για ε, το ποσοστό των θαλασσίων μεταφορών παγκοσμίω και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ακριβώς διεθνής από τη φύση τη αυτή ε, η ε, δραστηριότητα και θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ελκυστικότητα των θαλασσίων επαγγελμάτων. Το έχουμε ξανασυζητήσει επανειλημμένα για τα ναυτικά επαγγέλματα. Ο συνάδελφο Κουμουτσάκο μόλι είπε ε, ότι το κράτος σημαία είναι σημαντικότερο από το κράτος λιμένα, μα και τα δύο κράτη θα πρέπει να συνεργάζονται, να συμμετέχουν. Οι ε, συνθήκες εργασίας θα πρέπει να τηρούνται από όλους, γιατί μόνο έτσι θα είναι ελκυστικά αυτά τα επαγγέλματα και θα υπάρχει και ασφάλεια. Οι στόχοι μας, πώς να το πω, είναι τέτοια φύσεως ε, που είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Γι' αυτό το συζητούμε και το ε, κράτος λιμένα και μετά το κράτος σημαίες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι γενικά συμφωνώ με όλα ε, όσα είπε ο εισηγητής και βέβαια ε, θα πρέπει να έχουμε την ίδια διατύπωση παντού, ίσως και μεγαλύτερες προδιαγραφές. Ποτέ δεν θέλουμε να μην τηρούνται οι προδιαγραφές, βεβαίως ενημέρωση και πληροφόρηση που θα πρέπει να ε, διαβιβάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να είναι απόρριτες οι καταγγελίες και τα παράπονα, γιατί τα έχουμε ξαναζήσει, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται κανείς να ε, προσφεύγει, γιατί θέλουμε να μαθαίνουμε τα κακό σκήμενα, αλλά να προστατεύονται από εμπιστευτικότητα. Ο εισηγητής... Ε, επίσης αναφέρει και το θέμα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Πώς θα γίνει αυτό, συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να είναι επαόριστο. Ε, μετά από μία πενταετία, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει μια έκθεση ε, για να μπορεί κανείς να συγκρίνει. Μήπως χρειάζεται αναθεώρηση, έγινε κάτι που δεν έχει μπει στον κανονισμό. Δηλαδή, Ε, ε, προηγουμένως στο παρελθόν ήμουν ε, βουλευτή στην κάτω Σαξονία, στο τοπικό κοινοβούλιο. Περιοδικά κάναμε αναθεώρηση της νομοθεσίας για να βλέπουμε αν καλύπτονται όλες οι πτυχές, αν έχει προκύψει τίποτα καινούριο που δεν το έχουμε λάβει υπόψη. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι μεγάλη η ομοφωνία εδώ. Ο κύριος Τούσας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα που συζητάμε ε, για την ναυτιλία την ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή που αναφέρεται ουσιαστικά σε 1.200.000 ε, ε, εργαζόμενους. Ε, είναι πάρα πολλές οι γραφειοκρατικές οδηγίες, κανονισμοί, σε κοινοτικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται σε ζητήματα σε ό,τι αφορά τους όρους δουλειάς αμοιβή των αυτεργατών, αλλά και τους κανόνες ασφάλειας και αξιοπλοεία των πλοίων. Τι θέλω επιγραμματικά να αναφέρω. Ότι όλα αυτά, να μην είμαι απόλυτος, έχουν ελάχιστα αποτελέσματα θετικά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που οξύνονται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Με κύρια τάση ότι αυτό το βασικό πρόβλημα που έρχεται να λύσει η σχετική πρόταση όπως αναφέρθηκε εισηγητικά ότι δηλαδή δεν πρόκειται να χτυπηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά τους όρους δουλειάς αμοιβή των Ευρωπαίων αυτεργατών με αυτούς τους γενικούς κανόνες ε, έχω να παρατηρήσω το εξής. Τα ελάχιστα όρια που διαμορφώνονται σε ό,τι αφορά με τη Διεθνή Σύμβαση έχοντας υπόψη ε, πάρα πολύ σοβαρές τροποποιήσεις που έγιναν τα 20-25 τελευταία χρόνια θα πω στο επόμενο ζήτημα θα ασκήσουν και ασκούν όχι θα ασκήσουν ασκούν σοβαρή πίεση δίωξης χιλιάδων Ευρωπαίων ναυτεργατών με συγκροτημένα εργασιακά μισθολογικά δικαιώματα και αντικατάστασή τους με φτηνότερο ναυτεργατικό δυναμικό. Αυτή η τάση ε, εκφράζεται αν θέλετε στη χώρα μου με 124.000 ναυτεργάτες και 76.000 θέσεις εργασίας το 1978 και μιλάμε για το 2012 με τετραπλασιασμό του ελληνόχτητου στόλου με 24.000 περίπου 25.000 ναυτεργάτες και 16.000 θέσεις εργασίας. Εδώ ας μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτοί που έχουν αυτή την πρόταση στα ελληνικά πλοία στα αγγλικά πλοία, με σημαία αγγλική, με σημαία ελληνική, με σημαία γερμανική. Το πλήρωμα που θα είναι οι ναυτεργάτες που θα είναι με άλλες εθνικότητες θα έχουν τους όρους αμοιβή με βάση τη συλλογική σύμβαση της σημαίας που φέρνει το πλοίο ή με βάση τις διμερείς συμβάσεις που θα έχουν γίνει εκ των προτέρων μέσα από τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας. you, Mr. From the Commission. Ευχαριστώ. Κύριος Καραμίτσος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την έκθεση. Ε, ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Ε, όταν συζητήθηκε η σύμβαση αυτής της αρχές ε, του αιώνα και τελικά εγκρίθηκε το 2006 μετά πολλές προσπάθειες, ε, ανελήφθη δραστήριος ρόλος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για να συμμορφωθούν με τις διεθνείς αυτές απαιτήσεις. Στη συνέχεια, μεταγράφηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την ε, οδηγία 2006-2013. Όπως είπατε δεν ήταν με δεν ανήκει αυτό στην αρμοδιότητά μα, αλλά συζητήθηκε ανάμεσα στα συμβαλόμενα μέρη το ζήτημα τη παρακολούθηση και τη υλοποίηση. Τώρα συζητάμε το κράτο λιμένα και το κράτο σημαία. Ε, ήταν αναγκαία αυτή η συζήτηση για δύο λόγου. Πρώτον, για προχωρήσει η υλοποίηση τη νομοθεσία, διότι όπω σωστά είπατε, η Σύμβαση ναυτική εργασία ε, θα αρχίσει να ισχύει πλέον τον Αύγουστο το 2013 για τον τουρισμό, για την προστασία των ε, ναυτεργατών. Έσβησε το μικρόφωνο του μιλητή και δεν τον ακούμε ε, για να είναι πιο ελκυστικό το επάγγελμα και για την προστασία των αυτεργατών. Ε, κάτι άλλο που αναφέρατε και είναι εξίσου σημαντικό είναι η θεμητή όρη ανταγωνισμού. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το σύστημα, ούτω ώστε να μην εγκαταλείπουν τη Βρετανική ή την ελληνική σημαία ε, για να ε, βάλουν σημαία Παναμά. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η επιθεώρηση γίνεται πλήρω και ότι εφαρμόζονται όλε οι σχετικέ διατάξει χωρί καμία παρέκκληση. Στο παρελθόν έχουμε συζητήσει επί αυτό το θέμα με την ευκαιρία του Έρικα, του δικαστής και ε, το καθεξής. Πάντως, ε, στην νομοθεσία της Ένωσης, ε, τι γίνεται υλοποιεί το διεθνές δίκαιο, τα αποτελέσματα των διεθνών διαπραγματεύσεων και μεριμνούμε ώστε να υλοποιούνται αυτές οι διατάξεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συγκεκριμένα από τα κράτη-μέλη. Κοιτάζω τώρα τις τροπολογίες σας. Υπάρχουν 22 και τις περισσότερες μπορούμε να τις δεχτούμε. Ε, υπάρχουν και κάποιες που πρέπει να τις συζητήσουμε και μία που ε, σίγουρα έχουμε πρόβλημα ως θεσμικό όργανο για τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση. Αλλά αυτή είναι πάγια πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι έχουμε διάσταση απόψεων πάγια. Πάντως, πέρα από αυτό, εκκρεμούν και διάφορα άλλα ζητήματα που πρέπει να διευκρινίσουμε. Παραδείγματο χάρη το θέμα που αναφέρατε κι εσείς ε, η κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι αυστηρότερη σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις για κάποιες επιτυχές. Αληθεύει αυτό και εξακολουθούμε να είμαστε αυστηρότεροι από όλους και το θέμα ότι, έχουμε τον, ε, ότι θέτουμε επιτάπητος τον έλεγχο του κράτους λιμένα αυτό δεν σημαίνει ότι απεκδίονται κάποιοι άλλοι ευθύνε τους να εφαρμόζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος υπάρχει και το σοβαρό ζήτημα Τη κατάρτιση για όλους όσους ε, καλούνται να εφαρμόσουν τη σύμβαση. Οι αξιωματικοί ε, που λειτουργούν βάσει τη σύμβαση ναυτικής εργασίας ε, δεν είναι αξιωματικοί που θα αναλάβουν τις επιθεωρήσεις. πρέπει λοιπόν να σχετικοποιούμε τα ζητήματα. Εάν ε; μέσα στο παράρτημα, στον κατάλογο, Ε, τι τροπολογίε την 4 σχολιάσατε νομίζω. Αν ε, τέλο πάντων βάλουμε όλε αυτέ τι τροπολογίε στο παράρτημα τη οδηγία ε, για την MLC και αν πρέπει να εφαρμοστούν όλε αυτέ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ταυτόχρονα ότι δεν είναι ο σκοπό τη οδηγία στο παράρτημα. Υπάρχουν τίτλοι. Οι τίτλοι που υπάρχουν στο παράρτημα καλύπτουν τι συνθήκε εργασία. Σε βάση του μνημονίου του Παρισιού ανατίθεται στου αξιωματικού οι επιθεωρήσει, αλλά ε, προϊόν της διαδικασίας θα επανέλθουμε στο ζήτημα. Συμφωνούμε, όπω σα είπα, με τι περισσότερε τροπολογίε. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα ίσονο σημασία που θα πρέπει να διευκρινίσουμε, διότι μην ξεχνάτε ότι στο μέτρο του δυνατού ο στόχο μα ε, θα πρέπει να είναι να καταλήξουν συμφωνία τα δύο μέρη το συντομότερο δυνατόν δεδομένου το ότι το 2013 θα αρχίσει να εφαρμόζεται η σύμβαση, οπότε ιδανικά η οδηγία θα πρέπει επίση να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη, ώστε να γίνονται δεόντω οι επιθεωρήσει σε όλου του λιμένε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε σχέση με την ε, περίοδο τη μεταβατική πριν την υλοποίηση, 12 μήνη ή όχι, νομίζω τα μέρη θα πρέπει να το συζητήσουν αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαμίτσο, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Κουμουτσάκο, παρακαλώ να είστε σύντομο, ε, διότι έχουμε καθυστερήσει. Δύο δευτερόλεπτα, Πρόεδρο. Και στη βάση που οι πληροφορίε μου είναι σωστέ, ότι η Ελλάδα πριν δύο εβδομάδε κύρωσε ε, επίσης και εκείνη την MLC. Απλώ, επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριμένε χώρε, θα ήθελα να προσθέσω και αυτό στην λίστα των χωρών που την έχουν κυρώσει. Ευχαριστώ πολύ. states I read out were the ones... Τα κράτη που ανέφερε είναι αυτά που είχαν επικυρώσει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Έκτοτε επικύρωσε και η Ελλάδα, οπότε ναι. Ε, ουσιαστικά εγώ αναφερόμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έτσι ενημερωτικά τα ανέφερα όλα αυτά. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 16 Οκτωβρίου και στις 27 ε, Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και η Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα περάσει από την Ολομέλεια το ζήτημα. Έχουν διάφορε έχουν γίνονται διάφορε προβλέψει ε, για τι ε, ρογμέ ε, στην οροφή. Δεν ξέρουμε, τέλο πάντων αυτή είναι η αρχική πρόβλεψη. Και 16 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για τι τροπολογίε. Και περνάμε τώρα στην ευθύνη του Κράτου σημαία. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μα. Yes, Ο κύριο Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στη Συμφωνία του 2006 και ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, η ναυτική στον κόσμο είναι 1,2 εκατομμύρια. Ε, αυτό μπαίνει σε ένα συνολικό πακέτο. Ήδη ακούσαμε ένα τμήμα ε, για τη διεθνή ναυσιπλοεία και αυτό έχει να κάνει με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Λευκή Βίβλο ως εισηγητής καλωσορίζω εγώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα το θετικό αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι διατάξεις της συμφωνίας αυτή για την παρακολούθηση από το κράτος σημαία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση και πιο ε, σαφή. Και θα πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία αυτή και στα όσα ισχύουν για τον έλεγχο από τα κράτη σημαίες. Ε, για να μην έχουμε ε, αθέμητο ανταγωνισμό να προλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις. Όπως ε, θα είδατε από τη γνωμοδότησή μου, το κείμενο για την παρακολούθηση της στήρησης των ε, ρυθμίσεων το, έχω διευρύνει ε, και ε, ε, στις πιστοποιήσεις όπως προτείνει άλλωστε και η συμφωνία. Και επίσης έχω ε, αναφέρει τις επιθεωρήσεις και την εφαρμογή, την παρακολούθηση της υλοποίησης και της στήριξης των κανόνων, καθώς επίσης και ε, αρμόδιες αναγνωρισμένες αρχές και το προσωπικό τους και στο άρθρο 5 ε, η διαδικασία υποβολής παραπώνων και καταγγελιών στα πλοία. Αν θέλουμε να έχουμε ένα νέο σύστημα, αυτό είναι σημαντικό. Για το επόμενο διάστημα τώρα και τις ε, διαπραγματεύσεις και τις διαβουλεύσεις δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Νομίζω ε, το θέμα της πιστοποίησης και ερμηνεία του στα πλαίσια των νομικών αρμοδιοτήτων πρέπει να λυθεί. Ενδεχομένως ε, να μας απαντήσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι και περιμένω με χαρά τις προτάσεις των συναδέλφων και τη ε, συνεργασία με τους κοιόδες εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γιώργο και κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ζωσμπαχ, τον εισηγητή για το έργο του προηγουμένως είχα την ευκαιρία να πω ότι ακριβώς είναι αλληλένδετα αυτά τα θέματα. Και συνολικά καλό είναι που έχουμε μαζί αυτές τις προτάσεις και συζητούμε και το κράτος σημαίας και το κράτος λιμένα για να έχουμε ενιαίες ε, ε, συνθήκες εργασίας και για τους ναυτικούς. Δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι αυξάνει την ελκυστικότητα, την ασφάλεια αλλά και την ευρωπαϊκή ναυτιλία που θα αυξηθεί ε, έχει μεγάλη σημασία. Ε, θεωρώ πάρα πολύ σωστό και αυτό που λέει ο εισηγητής ε, για τη διατύπωση που την έχει προσαρμόσει στη Συμφωνία για την Αυτική Εργασία ε, και ε, αυτό ισχύει και για την προηγούμενη έκθεση, και τις αλλαγέ που προτείνει για την υλοποίηση και την εφαρμογή είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί συχνά χωλαίνει η υπόθεση. Και οι διαδικασίες καταγγελίας επί του πλοίου, όταν θέλει κανείς να υποβάλει ένα παράπονο, θα, ε, πρέπει να μπορεί να το κάνει παντού, ε, με διαφάνεια και με σωστέ διαδικασίε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο και χαίρομαι για τι συζητήσει που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Φλέκενστάιν, που ε, προεδρεύει στην Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας αυτή τη στιγμή και ε, λέγω το όσα θα σας έλεγε εκείνος. Ευχαριστεί τον εισηγητή για την γνωμοδότηση και καλωσορίζει την πρόταση που έχει κατατεθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση ε, με τη μορφή αυτή του ε, επιστοποιητικού και της δήλωσης ε, αξιοπλοείας για να εφαρμοστεί η ε, Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας. Επίσης θεωρεί ο κύριος Φλέκενστάιν, όπως και ο εισηγητής, ότι αυτή η πιστοποίηση θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και να υλοποιείται αυτό και να αναφέρεται ρητά στο διατακτικό, στα άρθρα. Γι' αυτό θα κάνει και τροπολογία ο κύριος Φλέκενστάιν, δεν την έχει υποβάλει ακόμα. Και τέλος, έχει και μια ερώτηση. Για ποιο λόγο η διαδικασία παραπώνων ή καταγγελίας επί του πλοίου που ήδη ε, ε, αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 13 του 2009. Γιατί επαναλαμβάνεται αυτό, αφού ήδη ρυθμίζεται αλλού. Ε, γενικά είναι θετική η γνωμοδότηση και πάλι ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τούσας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι ναυτεργάτες και το εργατικό κίνημα μέσα από αγώνες κατέκτησαν ορισμένα δικαιώματα που καταγράφονται στις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις εργασίας ανάλογα προφανώς με το συσχετισμό δύναμης. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπα προηγούμενα και ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, η αλλαγή των συσχετισμών δύναμης, η υποχώρηση του εργατικού κινήματος αντανακλάται και στο επίπεδο των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Ε, 38 συμβάσει ναυτική εργασία που εσωματώνονται στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 ε, υπονομεύουν ε, θεμελιώδη δικαιώματα των αυτεργατών. Χαρακτηριστικό σημείο, το πιο σοβαρό αρνητικό στοιχείο της ενοποιημένης Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας είναι η αναγνώριση ιδιωτικών υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και ναυτολόγηση των αυτεργατών που ουσιαστικά ενισχύει τον ρόλο των δουλεμπορικών γραφείων. Είναι πασίγνωστο, διεθνώς, όχι φυσικά μόνο στο πολιτικό επίπεδο στα στελέχη του ευρωπαϊκού Ευρωβουλευτές, στα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στους ναυτεργάτες, από άκρη από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική και Νότια Αμερική, ότι πλέον δραστηριοποιούνται ιδιωτικά γραφεία εύρης εργασίας που έναντι αντίτιμου χιλιάδων δολαρίων ο τζίρος τους είναι της τάξης των δισεκατομμύριων δολαρίων τα οποία εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο όπλων απομιζούν εκατομμύρια ποσά από τους λαθεργάτες αξιοποιώντας την αγωνία τους να βρουν δουλειά. Θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία αυτή και επιτρέψτε μου ένα σοβαρό γεγονός που έχει να κάνει με την εξέλιξη στη χώρα μας. Θα είμαι πολύ επιγραμματικός. Όπως διαπιστώνεται από τη σχετική ιστοσελίδα της φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα δημιούργησε ιδιωτικό γραφείο έδρασης εργασίας Ελλήνων στην έδεια. Αξιοποιεί αυτή η οργάνωση την αγωνία των ανέργων, επιτίθεται σε αλλοδαπούς και σε Έλληνες, απαιτώντας δουλειά για 12-14 ώρες με αμοιβή 18 ευρώ την ημέρα, με αλόγιστες συνέπειες. Οι εξελίξεις ό,τι αφορά την εφαρμογή της Γι' αυτό που προηγούμενα αναφέρθηκε για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα οι ναυτεργάτες να απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στον πλοίαρχο ε, καταστρατηγείται με τη διάταξη η οποία αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο που αναφέρει το εξή. Μπορεί να εφίσταται τιμωρία ο ναυτεργάτης που υπέβαλε καταγγελία η οποία έγινε προφανώς με οχληρό ή κακεντρεχή τρόπο. Δηλαδή, φτάσαμε σήμερα στο σημείο το ότι να ζητάει ο ναυτεργάτης να, του, εφαρμόζονται συλλογική σύμβαση εργασία, να καταβάλλονται οι δεδουλευμένοι του μισθοί, να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, οι συνθήκε, οι ανθρώπινε αξιοποιημένε συνθήκε δουλειά να μπαίνουν στο στόχαστρο ότι μπορεί πραγματικά να ζητεί κάτι με κακοκεντρή τρόπο. τέλος, επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγούμενα ότι είναι προφανές ότι αυτοί οι ελάχιστοι όροι που θεσμοθετούνται με τις τροποποιήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια θα ασκήσουν μεγάλη πίεση σε ό,τι αφορά στους ναυτεργάτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεμελιώδη μισθολογικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και γι' αυτό από αυτή τη σκοπιά εκφράζουμε την αντίθεσή μας. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καραμίτσος. Νομίζω ακόμα είμαστε στα θαλάσσια ύδατα, σε αλμυρό νερό, οπότε εσείς έχετε αρμοδιότητα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί πραγματικά μπήκε στο ψαχνό της υπόθεσης και εντόπισε κάποια πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Σίγουρα με κάποια επιμέρους σημεία μπορούμε να συμφωνήσουμε ο ρόλος των αναγνωρισμένων οργανισμών, εγκεκριμένων οργανισμών, με ποιο τρόπο θα πρέπει να χειρίζονται τις εμπλοκαταγγελίες. Ε, το θέμα της εμπιστευτικότητας είναι επίσης σημαντικό, αλλά το αναφέρατε και εσείς, Πρόεδρε. Όντως, όντως είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα και χαιρόμαστε που ε, με το έγγραφο επιφέρουμε βελτιώσεις ε, στο σύστημα. Ε, επίσης, ε, σε σχέση με τις διατάξεις για τις καταγγελίες, τις διατάξεις της MLC δηλαδή για τις καταγγελίες, ε, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χειρισμού, γιατί δεν αναφέρονται πολλά στην πρόταση αυτή. Άλλες πάλι διατάξεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας δεν αποτελούν τμήμα Τη κοινωνική συμφωνίες και κάποια σημεία είναι ευκολότερα. Η μισθή είναι δύσκολο σημείο, παραδείγματος χάρη, αλλά η ενδιέτηση και οι λεπτομέρειες ε, μπορούν να συζητηθούν, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιε κάποιες από τις διατάξεις προτείνει ο ε, να εξετάσουμε θα παρουσιάσουν ε, μικρότερη δυσκολία από άλλες. Αυτό ήθελα να πω. Και σε σχέση με το θέμα το πρώτο της πιστοποίησης. Δεν μπορούμε ή να το πω αλλιώ, υπάρχει ρήτρα πιστοποίηση μέσα στη Σύμβαση Ναυτική Εργασία, ε, δηλαδή το κράτο σημεία οφείλει να πιστοποιεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ζητήματα που δεν είναι αρμοδιότητα τη Ένωση, ε, π.χ. κάποιε κοινωνικέ πτυχέ ασφάλεια και, άλλες, ε, και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα μισθολογικά. Έχουμε λοιπόν την επιστοποίηση της ε, MLC, αυτό είναι ένα θέμα και ένα άλλο θέμα είναι αυτή η διάταξη. Τώρα το πώς θα το συνδυάσουμε δεν ξέρω γιατί θα δημιουργηθούν δυσκολίες, θα επικαλεστούν διοικητικές ε, δυσκολίες σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, εν πάση περιπτώσει, πριν από το επόμενο στάδιο, καλό θα ήταν να συζητήσουμε για να βρούμε κατάλληλες λύσεις, ε, χάρη στις οποίες θα εγκριθεί η πρόταση από τους συνομοθέτες ε, το ταχύτερο δυνατόν για να εφαρμοστεί και το ταχύτερο δυνατόν. Ε, ε, είναι θέμα πίεσης επίσης προς τα κράτη-μέλη για να κυρώσουν τη σύμβαση. Πίεσης προς τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη σύμβαση, ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει, γιατί και οι Έλληνες το άργησαν, το άργησαν, το έκαναν όμως. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για δημόσια κατανάλωση θα έλεγα ότι δεχόμαστε ότι η θαλάσσια πολιτική της Ένωσης δεν περιορίζεται στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, αλλά εντάξει, σίγουρα η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός παίκτη. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπάχα, έχετε τίποτα να προσθέσετε. Πάρα πολύ σύντομα μόνο. Γιατί ο συνάδελφος Ερτούκ με ρώτησε για ε, το άρθρο 5 της Συμφωνίας για την καταγγελία επί του πλοίου ε, για να υπάρξει αντιστοιχεία των κειμένων. Δηλαδή, να το λέει βέβαια η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, το λέει, αλλά θα πρέπει να το λένε και τα δικά μας κείμενα και να είναι η διατύπωση κάπως ενιαία για να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στα κείμενα. Αυτό μόνο. Γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαχ. Θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες για την έκθεση αυτή είναι επίσης 16 ε, Οκτωβρίου και ψηφίζουμε στις 27 Νοεμβρίου. 16 Οκτωβρίου τροπολογίες σας παρακαλώ. Ωραία. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της της διάταξης που είναι ε, στις 11 και 4. Ο παλιό φίλος ο Γιώργο Γερζεμπόφσκι είναι εδώ, εγκαίρος φυσικά και νωρίς ήρθε και θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα σε λίγο. Αν μας επιτρέπει, ε, ο ένα μικρό διάλειμμα για τον Πρόεδρο. Ναι, να κάνω και ένα τσιγάρο, λέει ο κύριος Γερζεμπόφσκι, που είναι γνωστός καπνιστής. Πέντε λεπτά διάλειμμα και αρχίζουμε. Colleagues, if you can take your seats again. Next item on the agenda is. Uh, Καθίστε, συνάδελφοι. Το θέμα της μερικής συζέταξης είναι η τριμηνιαία έκθεση του κυρίου Γιαζεμπόφσκι για το ΦΑΠΣ. για τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου. Όσοι ήθιστε να σου πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να σε βλέπω και πάλι εδώ στην Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών και έχεις το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Μπράιν, είναι δική μου η χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για τελευταία φορά για να σας αναφέρω την πρόοδο και την ε, μη πρόοδο όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα ενερίου χώρου ε, δύο μήνες πριν από την εκπνοή 4 Δεκεμβρίου 2012 ε, η γραπτή μου έκθεση έχει διανεμηθεί νομίζω ε, οπότε με τα χαρά θα απαντήσω τυχόν ερωτήσει στις λεπτομέρειες της διδαπτής έκθεσης και παρακαλώ να ακούσετε την σύνοψή μου. Καταρχήν θα ήθελα να διαφοροποιήσω την, πρώην, την τυπική μάλλον προ, ε, ε, καθιέρωση των ΦΑΜΣ και την ουσιαστική από την ουσιαστική. Για να σας ε, ενημερώσω για το τι συμβαίνει τύπης, ήμουν εδώ 24 Απριλίου, δύο κρατικές συμφωνίες έχουν συμφωνηθεί έκτοτε. Καταρχήν ε, για τον ΕΦΑ που είναι για τη Βόρεια Ευρώπη, Ιστονία, Λετωνία και Νορβηγία, Ιούνιο υπογράφει και αυτό και έπειτα Βαλτικό, Βαλτική ΦΑΜ, Λιθουανία, Πολωνία στις 17 Ιουλίου υπογράφηκε. Δύο ΦΑΜ λοιπόν και δύο λείπουν. Οπότε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε δύο μήνες πριν την εκπνοή της προθεσμίας ε, για να μην μιλήσω για τις εθνικές εποπτικές αρχές και τις σχετικές συμφωνίες και σε σχέση με τους παρόχους ε, υπηρεσιών αεροπλοείας ε, που πρέπει και αυτοί να συμφωνήσουν. Έχουμε το Blue Med Fab και μετά το Southwest Fab νοτιοδυτικό. Για το Blue Med θα θυμάστε ότι είναι η Ελλάδα στην ουσία και η Κύπρος. Έχουν ετοιμαστεί για την συνυπογραφή για τις 12 Οκτωβρίου. Τώρα την, ε, την ε, Παρασκευή μαζί με την διάσκεψη της ε, Λεμεσού για τον ενιαίο ουρά, ουράνιο χώρο. Και ποιον επισκέφθηκα για τον παλιό Υπουργό Μεταφορών της Ελλάδας, το συνάντησα την περασμένη εβδομάδα, τον Κώστα Χατζηδάκη που ήταν εδώ στην Επιτροπή μας πάρα πολλά χρόνια για την ε, νότιο-δυτική ΦΑΜΠΑ, την Πορτογαλία και Ισπανία δηλαδή, δεν ξέρουμε επισήμω πότε θα υπογραφεί. Κάπου λέει Οκτώβριο-Νοέμβριο μας λένε τυπικά. Ας δούμε, θα δούμε. Θα φανεί που λένε. Αυτά είναι τα τυπικά βέβαια. Αυτά που είναι πιο ενδιαφέροντα για εσά και για την πραγματικότητα, για του επιβάτε των αεροπλάνων, τι αεροπορικέ εταιρείε και τα αερολιμάνε είναι το τι έχει συμβεί ουσιαστικά. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι η στόχοι των λειτουργικών τμήματων εναερίου χώρου και η εγκαθίδρυση αυτών μέσα στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ήταν βελτιώσει στην, ε, στην ασφάλεια, στη χωρητικότητα, κόστος ωφέλεια και περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρότερες. Και να σας θυμίσω ότι τα εργαλεία για να τα πετύχουμε όλα αυτά μέσω των λειτουργικών τμήματων ανερίου χώρου είναι βασικά δύο. Ότι τα FABs θα πρέπει να φτάσουν μέσω της αναδιοργάνωσης του συστήματος ε, σε μια βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου και μια βέλτιστη χρήση ε, τεχνικών πόρων. Αυτά είναι τα υλικά για την ουσιαστική πρόοδο των FABs. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φτάνει την 1η Οκτωβρίου έκανε μια προσωρινή αξιολόγηση των πληροφοριών που είχε για τα FABs από τα κράτη-μέλη. Αυτή η προσωρινή αξιολόγηση θα ακολουθηθεί από μια επίσημη αξιολόγηση, την τελική, μετά από τις 4 Δεκεμβρίου. Ε, είναι εξαιρετική έκθεση και από όσο βλέπω Ό,τι και συμβεί μέχρι στου επόμενου δύο μήνες, το λυπηρό μου συμπέρασμα είναι ότι κανένα λειτουργικό τμήμα νερίου χώρου δεν θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει και στο βαθμό ανταπόκριση στις απαιτήσει, του όρου, θα απέχει πολύ. Όταν θα, αυτά θα δείτε στις λεπτομέρειες της έκθεσής μου. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχουμε εδώ τέσσερις κατηγορίες. Σχεδόν τέλειο εφαρμογή έχουμε μόνο στο δανέζικο ειδικό FAB. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον τα δύο εθνικά NSPs έχουν έχουν μετατραπεί, μεταμορφωθεί, γιατί αυτές οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι ένα κοινό NSP θα αναλάβει την λειτουργία αυτή. Αυτό που είναι παράξενο είναι ότι τα FABs και τα κριτήρια θα πρέπει να γίνονται άσχετα από τις, εθνικές, από τις χώρες και η Κομισιόν είπε ότι θα σκεφτόταν ότι θα ήταν καλό αν το δανέζικο σουηδικό ΦΑΜΠ συγχωνευόταν με το Ευρωπαϊκό ΦΑΜΠ. Θα θυμάστε ότι έχουν συνεργαστεί και έπειτα οι Δανείοι και η Σουδία φύγαν γιατί είπαν ότι οι άλλες χώρες είναι πολύ αργές για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ιδιών και έτσι ξεκίνησαν πολύ καλά και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι το δανέζικο-σουηδικό ΦΑΜΠ είναι σχεδόν τέλειο. Σχεδόν τέλεια εφαρμόγη. δεύτερη κατηγορία είναι αυτό που εγώ ονομάζω αρκετά καλά. Αρκετά καλή εφαρμογή Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Και, όχι, και γιατί δεν είναι καλύτερη από αρκετά καλή, γιατί έχουν κάνει πολλά με την καλή έννοια της διαχείρισης του εναέριου και τι δραστηριότητες που προσανατολίζονται στον ενέργειο χώρο, αλλά είναι κάτω από τις δυνατότητές τους όσον αφορά τον συνδυασμό και τη βέλτιστη χρήση των τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων. Εκεί έχουμε μείνει κάπω πίσω. Και το βλέπουμε και από την Κομισιόν που λέει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερη αποτελεσματικότητα αν ήθελε. θα πρέπει να δούμε ότι όλες οι διατλαντικές και υπερατλαντικές ε, πτήσεις που περνάνε, φεύγουν μάλλον από το κέντρο της Ευρώπης περνάνε από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την ε, Ιρλανδία. Εκεί υπάρχει χώρος για βελτίωση. Τρία. Μερική εφαρμογή, το ονομάζω εγώ. Ποιες χώρες είναι εκεί, ποιο, ποιο φάμιλα, του Δόναβη και του Ισβαλτικής. Το ΦΑΜ του Δούναβη, Βουλγαρία και Ρουμανία δηλαδή έχουν ξεκινήσει καθυστερημένα αλλά προσπαθούν να κάνουν πρακτικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση του νερίου χώρου. Το βαλτικό ΦΑΜΠ ε, ήταν πολύ καθυστερημένο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι χώρες που μπορούν να συνεργαστούν. Και τα δύο ΦΑΜΠ είναι, είναι ε, με δύο χώρες και είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν δύο χώρες. Αλλά για να είμαστε ειλικρινή το βαλτικό φαμπ είναι ε, μάλλον σε χειρότερη κατάσταση. Γιατί έχουμε και λίγη Πολωνία και λίγη Λιθουανία μέσα. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούν να συγχωνευτούν με άλλα φαμπ. Τέταρτη κατηγορία μου είναι πέντε φαμπ δυστυχώς, όπου θα έλεγα ότι η εφαρμογή απουσιάζει. πολύ λυπηρή εξέλιξη και θα θυμάστε το Φαμπέκ. Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και κτλ. Πολύ απογοητευτικά όλα αυτά γιατί πέγραψαν την κρατική συμφωνία το 2010. Δύο χρόνια δηλαδή μετά την υπογραφή δεν έχει γίνει καμιά κίνηση. Το μεγαλύτερο φαμπ τώρα είναι το 55% των νερίου χώρου μας είναι αυτό. Χρειάζεται να γίνει πρόοδος εδώ. Βέβαια, οι έξι χώρες έχουν κάποιες ιδεολογικές διαφορές, όπως τα γνωρίζετε, και από τους ε, σιδηροδρόμους. Ελαφρές διαφορές στην ιδεολογία και στις αντιλήψεις τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι το ΦΑΜΠΕΚ θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με τους ε, οι θύνοντες έγινε μια μεγάλη συνάντηση πέρσι και υποσχέθηκαν κάτι προγράμματα εργασίας ώστε σταδιακά να βελτιωθεί η συνεργασία και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα κτλ. κτλ. φέτος το καλοκαίρι ξανασυναντήθηκαν στο Λέβεν και έχουν και πορίσματα του Λέβεν, αλλά στην πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα πρόγραμμα εργασίας ε, για να αναζητήσουν ε, τις δυνατότητες βελτίωσης. Αλλά όπως σας είπα, δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα, το Fabs CE. Δεν θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη Αυστριακή Αυτοκρατορία, αλλά είναι σχεδόν ε, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κροατία κτλ. Και εδώ τα ίδια συμβαίνουν. Πολύ δύσκολο 7 χώρες να φτάσουν σε συμπεράσματα μέλη ήταν ελεύθερα να διαλέξουν τι είδους φαμπ θέλαν να φτιάξουν. Είχαν απόλυτη ελευθερία. Και τα αποφασίσαν από τον Μάιο του 11. 1,5 χρόνο πριν δηλαδή περίπου. Είχαν αρκετό χρόνο νομίζω. Τα υπόλοιπα τρία είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά είναι σημαντικά. Είπα ήδη για τον Νίφαμπ. Το Νίφαμπ άργησε να ξεκινήσει και είναι λίγο ενοχλητικό ότι η εφαρμογή για την νεότερη συνεργασία δεν έχει στόχο το 2012, αλλά το 2015. Δεν είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα που υποτίθεται ότι θα είχαν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έχουν ξεκινήσει. Και Υπάρχει, έχουν και την Νορβηγία στο σύστημα που είναι σημαντικό. Για το νοτιοδυτικό ΦΑΜΠ πολύ απογοητευτικό γιατί ξεκίνησε νωρί. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν κάνει υπογράψει την κρατική του συμφωνία. Το καλοκαίρι ήμουν στην Ισπανία και την άνοιξε στην Πορτογαλία. Εντάξει, υπήρχαν και εκλογέ, νέα, κυβέρνηση στην Πορτογαλία κτλ. Αλλά νομίζω πως ε, δεν είναι, είναι εύκολο το ΦΑΜ αυτό για διοργάνωση και ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρώσουν την ε, συμφωνία. Το πιο δύσκολο είναι το Blue Med, γιατί οι πολιτικές και οι οικονομικές δυσκολίες ε, της Ελλάδας και της Κύπρου είναι πασίγνωστες, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία γιατί η νομοθεσία αυτή χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2009 και τρία σε τρία χρόνια θα έπρεπε να είχαν κάνει κάποια πρόοδο για να επιτύχουν τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου και των τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων στα δύο επίπεδα NSP και NSA. Ποιε είναι λοιπόν οι ιδέες μου για το μέλλον. Να σας δώσω τέσσερις ιδέες, προσωπικές ιδέες Εγώ νομίζω πως θα ήταν θετικό αυτή η Επιτροπή να στείλει σαφές μήνυμα στα κρατημέλη και ε, διάβασα και την έκθεση Φώστερ ξανά το Σαββατοκύριακο. Είναι καλή έκθεση αυτή και αξίζει ε, καλής μεταχείρισης τον Οκτώβριο εδώ στο Κοινοβούλιο. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να πούμε επιταχύνεται την, ε, τα όσα πρέπει να κάνετε. Εμείς σας στηρίζουμε. Σας στηρίζουμε, θα πρέπει να ξεκινήσετε τις απαραίτητες κατά παράβαση διαδικασίες αμέσως από το 2013, γιατί είναι σαφές και νομίζω πως κάποια πράγματα παραπάνω θα τα μάθουμε από τις ιδέες, για τις ιδέες του Κομισιόν μέσω της ομιλίας του Αντιπροέδρου Κάλλας που στη Λεμεσό την Πέμπτη. Ο Πρόεδρος σας θα είναι εκεί, θα κάνει και εκείνος μια ομιλία. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ε, είναι πολύ σημαντικό να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν. Γιατί η νομοθεσία φτιάχτηκε το 9 με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρία χρόνια έπρεπε να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί αυτά όλα τα κάνουμε για την οικονομία και για το περιβάλλον της Ευρώπης. Θέλουμε να υπάρξει βελτίωση της ασφάλειας, ε, αύξηση της χωρητικότητας και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η δεύτερη μου άποψη είναι κάτι που όλοι το θέλουν, αλλά νομίζω πως θα πρέπει κανείς ε, να υποστηρίξει μια την ε, διπλή προσέγγιση για το FabCE και το FABEC. Γιατί άμα περιμένουμε μέχρι η Βοσνία να βρει άκρη και για το FABEC βέβαια ισχύει αυτό, αν σε τρία χρόνια δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν σε συμπέρασμα μαζί, ε, τότε θα πρέπει κανείς να αρχίσει μια προσέγγιση δυο ταχυτήτων. Έχουμε, κάνει, έχουμε καλά παραδείγματα. Σκεφτείτε το Schengen, το Eurogroup, Κάποιοι θέλουν να κάνουν αυτά που είναι απαραίτητα και να τα κάνουν ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να μπουν αργότερα. Γιατί διαφορετικά, αν περιμένουμε μέχρι να συμφωνήσουν 6-7 χώρες για ένα πρόγραμμα, δεν θα σημειωθεί η πρόοδος. Τι είναι το μήνυμα. Είναι απαραίτητο να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και να τους πούμε ότι θα πρέπει να κάνουν προσκλήσεις στα υπόλοιπα μέλη για να μπουν στα FABs. Ένα πολύ σημαντικό είναι η Ισλανδία που είναι υποχρεωμένη στην ουσία να μπει στα ΦΑΜΠ γιατί σύμφωνα με τους, ε, τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι υποχρεωμένη να μεταγράψει την νομοθεσία ECS στην εθνική της νομοθεσία και μετά να μπει σε ένα ΦΑΜΠ. Και στην ουσία κάνουν πλάκα αυτοί. Πριν από κάποιους μήνες ήμουν στην Ισλανδία και ο υπουργό είπε ε, ναι, ξέρεις ότι το κόμμα μου δεν είναι υπέρ του να γίνουμε μέλος, αλλά εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τώρα πρέπει πια να κάτι να κάνουν. Πάντως, αυτό που είναι πιο πολύ σημαντικό είναι τα υπόλοιπα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Να δείτε την τελευταία σελίδα της εκθεσής μου, θα δείτε ότι στο B έχουμε την Αλβανία, τη Μακεδονία, το Μοντενέγρο, Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Θα δείτε δε στο χάρτη στην πρώτη σελίδα της εκθεσής μου ότι είναι μέσα στον εναέριό μας χώρο. Άρα θα ήταν λογικό να καλέσουμε τις χώρες αυτές να μπουν στα ΦΑΜΠ. Γίνονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά από όσο γνωρίζω δεν έχει υπάρξει ποτέ γραπτή πρόσκληση προς τις χώρες αυτές. Τέσσερα. Θα πρέπει προσεκτικά να αναλύσουμε την κατάσταση και να σκεφτούμε νέε πρωτοβουλίε συμπεριλαμβανομένε τη ε, πιθανή ε, τροποποίηση τη νομοθεσία ECS. Ε Κατά τη γνώμη μου αυτό μπορεί να γίνει με τέσσερις τρόπου. Ορισμένα φάβες έρχονται και λένε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το NSP γιατί υπάρχουν διαφορετικές ε, διαφορετικές ε, πολιτικές και καθεστώτα. Θα πρέπει, νομίζω πως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις εθνικές υποχρεώσεις για να διευκολύνουμε τα FABs. Έπειτα θα πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για τα FAB, για τα κοινά τεχνικό σύστημα. Πρέπει να βελτιώσουμε τα διασύνδεση ανάμεσα στα FAB και τη συνεργασία μεταξύ αυτών. Και το 4, και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι και μείωση των FAB μέσω συγχώνευσης. Το τέσσερα είναι και αυτό είναι που λέει ο Πίτερ, ε, έρθει, να έχουμε δεσμευτικούς στόχους για την επόμενη περίοδο. Να πιέσουμε τα, πιέσουμε τα κράτη, να ότι δεν θέλουμε μόνο την οργάνωση, θέλουμε και τα αποτελέσματα. Mm. Τώρα, ο συντονιστής του Ζουσουφάμπ από την, ε, την ε, νομοθεσία SS, SES, ε, e ο διορισμός μου εκπνέει, θα ήθελα ωστόσο να ευχαριστήσω καταρχήν την Κομισιόν ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά να στηρίξω αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας των ΦΑΜΠ και να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Κάλλας και το επιτελείο του καθώς και τους υπαλλήλους της DG Move μου για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη δουλειά και για τη στήριξη που μου ε, προσέφεραν. Και επειδή το έργο μου στηρίχθηκε πάρα πολύ από αυτήν την Επιτροπή, πράγμα που βοήθησε όταν πήγα στις πρωτεύουσες κάποιων χωρών για να τους πιέσω ε, λέγοντας ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει αυτή την ιδέα, λέγοντας λοιπόν ότι αφού ε, με στηρίξατε θα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, του συντονιστές και τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, George. I think we should thank you as well. Σε ευχαριστούμε, George. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς γιατί ήταν δύσκολο το έργο σου και δύσκολες και οι συνθήκες τι οποίο το επιτέλεσε. Άσε που είχες ε, παρεδώσει με πολύ δύσκολους ανθρώπους από τα κράτη-μέλη. Ε, ένας λιγότερο αποφασισμένος ή όχι τόσο ικανός θα τα έχει εγκαταλείψει ήδη. Ο αντιπρόεδρος Κάλλας σκεφτόταν, ε, όταν σκεφτόταν να στο αναθέσει, του είπα εγώ ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο γιατί είναι αποφασιστικό ο Τζορτ και επίμονο και τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται όταν μιλάμε για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Δεν έχουμε ακόμη τέτοια blogs και θα δεχτούν όλοι ότι χρειάζεται χρόνος για τα θαύματα. Αλλά πάντως ε, και εδώ που έχει στάσει, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. προλύανε στο έδαφος για τις μελλοντικέ εξελίξεις. Σε σχέση με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου που ζητάς, εγώ θα περιμένω το Simpson, ε, θα περιμένω εγώ προσωπικά την ομιλία την πέμπτη το πρωί και νομίζω καταλαβαίνεις γιατί τηρώ τέτοια διπλωματική στάση. <laughs> θα τα πούμε την πέμπτη το πρωί. Ευχαριστούμε, Μάτιο. Ματιό ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τον συνάδελφό μας τον Γεώργ Γκέρτζαμπόφσκι. Δυστυχώς, οι διάφοροι φόβοι επαληθεύτηκαν τους τελευταίους μήνες. Τώρα βρισκόμαστε και σε μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια. Τα έχει ζήσει εσύ πάρα πολύ συχνά το Συμβούλιο υπογράφει διάφορα πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζονται. Αυτή είναι η παλιά πληγή. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να πούμε στο Συμβούλιο και να το πιστέψει ότι δεν μπορεί από τη μια διαρκώς να διαπιστώνει ότι οι πολίτες στην Ευρώπη δεν πιστεύουν ουσιαστικά στην Ευρώπη εάν δεν είναι σε θέση το Συμβούλιο να εφαρμόζει τα όσα αποφασίζει το ίδιο σε τόσο σημαντικά θέματα όπως αυτά εδώ που είναι θέματα ασφαλείας. Ε, ε, είναι όλοι ε, διάπηροι με λάβαρα και μετά και όταν πρόκειται να εξοικονομήσουμε και χρήματα, όλα αυτά απασχολούν όλες τις κυβερνήσεις. έχουμε ένα σχέδιο τώρα, καλούνται να το εφαρμόσουν, δεν το πράττουν. Γι' αυτό θεωρούμε εμείς από το ΕΛΚ ότι θα ήταν πάρα πολύ λάθος μήνυμα ε, να κάνουμε τις βαλίτσες μας τώρα, να εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια και να προσπαθήσουμε να φέρουμε νέα νομοθεσία. Όχι. Νομοθεσία υπάρχει. Χωράει βελτιώσει. Αλλά να δείξουμε στι χώρε ότι δεν είναι αυτή η συμπεριφορά, ούτε μπορούν να παίζουν με το κοινοβούλιο, ούτε με του πολίτε του. Κατά τα άλλα, την ιδέα των δύο ταχυτήτων τη θεωρώ πολύ σωστή. Δηλαδή, εκείνοι που θέλουν να κάνουν ένα πιο ταχύτερο βηματισμό να έχουν την ευκαιρία στο ίδιο λειτουργικό τμήμα εναριού χώρου και αυτό θα ε, λειτουργήσει και με πιστικό τρόπο για να οθήσει και τους υπολείπους να ακολουθήσουν ε, και να κινητοποιήσουν τα θετικά τους αντανακλαστικά. Ε, λέω λοιπόν ρητά ότι δεν θέλουμε νέα νομοθεσία και κανονικά θα, θα προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην τα αγγίξει όλα αυτά και ανταυτού ε, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της όταν δεν υλοποιούνται οι νομοθεσίες. Ένα άλλο θέμα. Τώρα αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα σαφές μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι στάση αναμονής. Για να δούμε και ελπίζω ε, την ομιλία που θα εκφωνήσεις Μπράιαν εσύ και ο Επίτροπος να πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Και κατά την άποψή μου αυτό το κεφάλαιο δεν θα πρέπει να το κλείσουμε με μια ελπίδα να κινηθεί κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Δεν πρόκειται να κινηθεί εάν δεν πέσει ράβδος και εγώ πραγματικά θα ήμουν υπέρ αυτής της οδού. Ένα τελευταίο, δηλαδή τώρα είναι το πραγματικό τελευταίο, τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου. Ξέρουμε τις δυσκολίες ε, και θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ε, μία από τις δυσκολίες έχει να κάνει με το καθεστώς των ανθρώπων που εργάζονται αυτό το καιρό. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και με τον Ζόρς Μπαχ. Πρέπει να, να βγούμε από αυτές τις αγγυλώσεις, τις διαδικαστικές. Να μην ε, επιβάλλουμε τη μία ή την άλλη επιλογή, αλλά την καλύτερη δυνατή λύση εντός ενός λειτουργικού τμήματος. Το πρόβλημα εκεί θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, εκεί που χωλαίνει και να πούμε ότι δεν είναι δικός μας ρόλος να προτείνουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, να τα βρούνε μόνοι τους. Οι συμφωνίες διακρατικές είναι. Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ε, για την σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Ο κύριος Ελχαντράουι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γκέαρκ για την εισαγωγή του και για όλη τη δουλειά αυτή που έβγαλε σε πέρα στο τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι παρά τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί εδώ και εκεί, ε, στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Οι στόχοι της νομοθεσίας. Και σίγουρα δεν υπάρχει ε, πραγματικά λειτουργική εφαρμογή των FAPS με το μεγάλο δυναμικό που γνωρίζουμε όλοι. Θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος τώρα για το τι μέλη γενέστε. Πώς ε, θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Η μπάλα βέβαια είναι τώρα στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα έλεγα όπως ήδη είπε ο Ματιο Γκρός, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα τι πρόκειται να κάνει. Ε, δεν υλοποιείται η ε, νομοθεσία, πρέπει να επιβάλλει την εφαρμογή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις νομικές τους και νομοθετικές υποχρεώσεις. Συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Γιαζεμπόφσκη όταν λέει ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να προχωρήσουν και άλλες να μην προχωρήσουν. Ε, ε, να μην παρεμποδίζονται λοιπόν εκείνες που θέλουν να προοδεύσουν από τις υπόλοιπες. Συμφωνώ με αυτό, να δούμε πώς θα το οργανώσουμε πρακτικά. Το σημαντικότερο είναι να έχουμε στην πράξη αποτελέσματα. Ένα επόμενο σημείο, τρίτο που πρέπει να συζητήσουμε ίσως με τους συντονιστές, Μπράιεν. είναι επειδή έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, μήπως θα είχε νόημα να συστήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει ε, τη θητεία του κυρίου Γιάρτζεμπόφσκι. Δεν ξέρω αν το επιθυμεί ο ίδιος. Ε, γιατί ε, το Δεκέμβριο δεν θα έχει λυθεί αυτό το θέμα, δεν θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί επειδή είναι συντονιστής και τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα, μπορεί να μας ενημερώνει και στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, να κοιτάξουμε ε, πώς θα γίνει αυτό με την εντολή, αν μπορεί να παραταθεί η θητεία του. Νομίζω ότι ο κύριος Γιάρτζεμπόφσκι θα πρέπει να έχει ε, αρκετές εξουσίες για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό ήθελα να προτείνω. Αν δεν διαφωνούν συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι καλό. Τον ίδιο τον Γκέορκ, θέλω να το ρωτήσω κάτι για το Φαμπέκ. Ποιο είναι τώρα το μεγαλύτερο εμπόδιο και ο μεγαλύτερο σκόπελος. Γιατί αν υλοποιηθεί το Φαμπέκ είναι ε, η μισή ενέργεια κυκλοφορία, το 55%. Λοιπόν, ποια είναι τα εμπόδια εκεί, πού σκοντά αυτή η υπόθεση, πώς μπορεί να λυθεί και ε, έχετε και εκεί την ίδια πρόταση να προχωρήσουν ορισμένες χώρες ενώ κάποιες άλλες δεν προχωρούν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάισνε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γιάννη για την παρουσίασή του. Στην αρχή ακούστηκε πάρα πολύ πιστικός και αποφασιστικός και μετά είδαμε ποια είναι τα προβλήματα. Μα είναι τρελά πράγματα αυτά. Συμφωνώ με το Μάτιο. Πολλά πράγματα υπογράφονται, αποφασίζονται και κανείς δεν ε, τα εφαρμόζει. Το έχουμε και στον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό και στο πακέτο για το σιδηρόδρομο. Καμιά φορά δεν αξίζει τίποτα ούτε καν το μελάνι για τα χαρτιά στα οποία είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα. Γενικά το καταλαβαίνω στις ρυθμίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στο κάτω-κάτω είναι και θεματοφύλακα των συνθήκων ε, θέλει να έρχεται και να εφαρμόζει εκείνη διάφορα και να έχει την εκτελεστική εξουσία και, και ε, Εμεί αυτό δεν το θέλουμε στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει επικουρικότητα και μπορεί κανεί να προσφεύγει και στο δικαστήριο. Αλλά τώρα ε, κανονικά όλοι οι πολίτες θεωρούν ότι τα αεροπλάνα στην Ευρώπη κυκλοφορούν ε, όπως δείχνουν ε, αυτά τα ωραία περιοδικά που έχουν τα αεροπλάνα που δείχνουν τη σύνδεση των αεροδρομίων σε ευθεία γραμμή. δεν γίνεται όμως έτσι και τα κράτη-μέλη ακριβώς και μόνο εντός της Ευρώπης δεν μπορούν σε αυτά τα μικρά κομματάκια του πάζελ να τα συντονίσουν, γιατί δεν μιλάμε καν για ε, ένα αέριο χώρο ενιαίο. Μιλάμε για λειτουργικά τμήματα. Αυτά τι είναι ψηφίδε. Ούτε αυτά δεν μπορούν να φτιάξουν. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Και άντε να το εξηγήσει αυτό στον πολίτη. Ε, ε, τι μπορεί να γίνει. Μπορούμε να πούμε να λάβει τις ευθύνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λόγω της μη εφαρμογής. Ναι, αλλά αυτό δεν νομίζω να εφαρμοστεί. Ε, και συμφωνώ με τον Σαΐντ να ανανεώσουμε τη θητεία. Γιατί αν πούμε ότι είχαμε ένα συντονιστή, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, ο, άνθρωπος ε, προσπάθησε, αλλά τι να κάνουμε. Μα αυτό είναι και τελικά υπόθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον κάτι δεν εφαρμόζεται, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό με τι δύο ταχύτητε. Καλή πρόταση είναι, αλλά για το ΦΑΜΠΕΚ, γιατί εμεί οι τρει που μιλήσαμε από τη ΦΑΜΠΕΚ είμαστε, πώ θα λειτουργήσει αυτό, γιατί ε, που χωλαίνει στου δύο μεγάλου, Γερμανία ε, και Γαλλία, που έχουν τάξει λαγού με πετραχίλια και δεν τα εφαρμόζουν γιατί το συζήτησα με τους Γερμανούς και λένε οι Γερμανοί εμείς έχουμε το καλύτερο σύστημα να προσαρμοστούν οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι σου λένε σιγά μην προσαρμοστώ, να προσαρμοστούν οι Γερμανοί στο δικό μου σύστημα. Ε, και τώρα πώς υπάρχει εξασφάλιση πτήσεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας ε, χωρίς να ρίξουν τα μούτρα του στα κρατη για να προσαρμοστεί ο ένας στον άλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ και τον πρώην συνάδελφο για την ωραία του έκθεση. Έχω μια μικρή επιθυμία κύριε Γιάννη και παράκληση. Όταν μιλάτε για ΦΑΠΤΕ, μη λέτε παλιά Αυστρία, Αυστρο-Ουγγαρία ή Αυστριακή Αυτοκρατορία. Μα γι' αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί ακριβώς τέτοια αποθυμένα έχουν όλοι από αυτές τις εποχές. Και δεν ξέρω κανέναν από εκεί. Παρακαλώ, μην κάνετε τέτοιες αναφορές. Ε, πάντως, είναι ε, ε, υποδειγματική η κατάσταση. Αυτή η FAB, αυτό το λειτουργικό τμήμα, το FAB C, περιλαμβάνει πολλές μικρές χώρες. Και ε, γι' αυτό είναι ακόμα πιο επίγον το συντομότερο να συνεργαστούν πιο συχνά και πιο στενά. Γιατί αυτή ήταν και η πρόθεση. Πολύ μικρή μαζί να κάνουν μια μεγάλη ενότητα. Από ό,τι φαίνεται απέτυχε εκτρά αυτή η προσπάθεια. Και σας ερωτώ, ποια είναι εδώ τα πολύ μεγάλα εμπόδια. Γιατί είναι πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή βέβαια, αλλά υπάρχουν και χώρες εκεί που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά όμως, ακούω ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι και τελείως απρόσκοπτη η συνεργασία ήδη δηλαδή των κρατών μελών μεταξύ τους. Και έχω και μια ερώτηση για ε, την πολεμική αεροπορία που έχει αποκλειστικότητα σε κάποια κομμάτια του εναέριου χώρου και απαγόρευση για τις ε, πολιτικές πτήσεις. Πώς έχει εξελιχθεί αυτό το θέμα. Νομίζω είναι θετική και ευνοϊκή. Και να ρωτήσω κάτι για το νότιο-ανατολικό ε, μεσογειακό. Να το δυτικό εννοεί ο Μιλήτρια γιατί ρωτάει για το Γιβραλτάρ. Υπάρχει ακόμα αυτό το πρόβλημα με το Γιβραλτάρ. <laughs> Γιατί αυτό είναι ένα θέμα λίγο που επανέρχεται σαν παλιό τροπάρι, σαν ένα φάντασμα ξανά. Μόλις πεις τίποτα για ένα αέριο χώρο πετάγεται το Γιβραλτάρι. Παρόλες τι επιφυλάξεις της κυρίας Μάισνερ, ε, να συζητήσουμε για την ανανέωση της θητείας εγώ κατάλαβα ότι είπατε εμεί θέλουμε κανένα λάθο μήνυμα. Ναι, το κατάλαβα λάθο, γιατί εγώ έτσι το εξέλαβα, να μην ανανεωθεί η θητεία. Όχι, όχι, να ανανεωθεί. Γερμανικά τα είπα. νομίζω πρέπει να διατηρηθεί η πίεση και να το λύσουμε αυτό το θέμα, Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτούς τους εθνικούς εγωισμούς. Αυτό είναι το ζήτημα ε, σε αυτή την ιστορία. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουν ότι ε, δεν έχουν την πανάκια ή το απάβγασμα ε, του μοντέλου η κάθε χώρα. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τελικά θα καταλήξουμε να έχουμε μόνο ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών πολιτικής αεροπορίας. Ε, τότε Το έχει ξαναπεί και ο Σέξπιρ αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα, είναι μια τρύπα στο νερό και μια μάταιη αγάπη. Ο κύριος Κράμερ. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντα όταν βλέπω τον κύριο Γιαρτσεμπόφσκι και εδώ δεν διαφωνούμε και δεν μπορούμε καν να τσακωθούμε. Άκουσον, άκουσον. Ε, ε, πώς αλλάζουν οι καιροί. Πού να το έλεγε κανείς. Αλλά το είχα πει από την αρχή ότι για αυτή τη δουλειά είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και γι' αυτό ε, θέλουμε να παραταθεί η θητεία του, τα πρότεινε και η Γκεζίνε. Αλλά είναι τρελή η κατάσταση. Αυξάνεται η ασφάλεια, αυξάνεται οι οικονομίε, προστατεύεται το περιβάλλον. Αυτή είναι η πρωτογενή στόχη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συμφωνήσει οι πάντε, ομόφωνα. Και δεν εφαρμόζεται. Ακούστηκε η Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι έχουν οικονομικά προβλήματα. Ε, ναι, το έχει καταλάβει μέχρι και η Ελλάδα αυτό αλλά ε, ότι να υπάρχουν αντιστάσεις παρόλο που μπορούμε να κάνουμε εδώ οικονομίες χωρίς να πλήττονται οι φτωχοί, χωρίς να είναι μεγαλύτερη καταστροφή, χωρίς να αυξάνεται ο ΦΠΑ. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν προχωρούν. Ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Όλοι θέλουν οικονομίες, όλοι θέλουν λεφτά, όλοι έχουν οικονομικά προβλήματα και εκεί μπορούν να το λύσουν κομψά, μόνο με πλεονεκτήματα μην το κάνουν. Και θα με ενδιέφερε, ε, στις συζητήσεις αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Όταν λένε διάφορες χώρες δεν μπορούμε, η απάντηση ποια είναι. Ε, πώς θα σωθείτε από την οικονομική κρίση, πώς θα εξοικονομήσετε χρήματα. Εκεί μπορούμε να συνέσουμε και τους τρεις στόχους. Ε, θα ήθελα περισσότερα επιχειρήματα. Πώς απαντούν ανερυθρίαστα. Πώς τολμάνε και ανοίγουν το στόμα τους. Εδώ και τρία χρόνια. Ξέρετε πόσα λεφτά θα είχατε εξοικονομήσει. Εφαρμόστε το επιτέλους. Thank you, πριν ξαναδώσω το λόγο στον Τζορτ και στην Επιτροπή, να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Απήχω άλλε παρεμβάσει βέβαια. Ξέρω ότι Δευτέρα θα συζητήσετε άμεσα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο λόγους. Πρώτον, δεν έχει γίνει η δουλειά, δεν έχει ολοκληρωθεί, όχι ότι τη εσύ. Και δεύτερον, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο για να γίνει τελικά η δουλειά. Είναι σημαντικό. Για να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους υπουργούς. Ε, δεν ξέρω ακριβώς τι με περιμένει κάθε φορά που μιλάω με τους υπουργούς. 25 χρόνια σχεδόν έχω εδώ στο Κοινοβούλιο ε, και δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο δόλιο συμβούλιο όπως ε, το τωρινό. Και όχι μόνο για αυτά, αυτά τα λειτουργικά τμήματα ένα αερίου χώρου, αλλά για όλα τα ζητήματα μεταφορών. Μια σειρά ζητημάτων υποσχέθηκε το Συμβούλιο, υπέγραψε, Έδωσαν το λόγο τους και τίποτα δεν κάναν, τίποτα απολύτως. Ε, ο Κρόμβολ, όταν το ρώτησαν για τον Κάρολο, το πρώτο που είχε υποσχεθεί ότι θα αναθεωρήσει το καταστατικό του κοινοβουλίου, ε, ε είπε λοιπόν ότι είναι ε, σαν... Ε, είναι πάρα πολύ εύθρυπτες οι υποσχέσεις του, του Καρόλου. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και εγώ για το Συμβούλιο. Δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να τους πούμε. Ό,τι και αν θέλετε να κάνετε με την τωρινή Προεδρία, εμείς ε, δεν σας εμπιστευόμαστε. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σχέσεις μας με το Συμβούλιο για αυτό το τομέα. Ε, και όταν μιλάω και με τους υπολείπους μου λένε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δικό μας ε, το τομέα. μας κάνουν κηρύγματα για τον προϋπολογισμό ε, και μας λένε ότι χρειαζόμαστε περικοπές 150 εκατομμυρίων ευρώ, λιρών, τέλος πάντων οτιδήποτε. Αλλά αν εκείνοι φύρμοζαν αυτά που, τα, τα υπεσχημένα, θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν όχι μόνο εκατομμύρια, να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης και ανταυτού τίποτα. Μηδέν, δεν έχουμε κάνει τίποτα και κρύβονται πίσω από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το 89 λέγουν κάποιοι ότι με την κατάρρευση του τείχους άνοιξε η Ευρώπη. Συγγνώμη ότι ε, ανταυτού έχουμε 27 τείχη του Βερολίνου ε, που έχουν ορθώσει τα κράτη-μέλη για τον εναέριο χώρο. Και λέω, στρεφόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέα νομοθεσία, όχι, όχι, λέμε όχι. Φτάνει. Είναι μια χαρά αυτή η νομοθεσία. Πότε ήταν Τζόρις που έπρεπε να είχαν υπογράψει όλοι. Στις 4 Δεκεμβρίου, στις 5 στις 4 Δεκεμβρίου 2012 η ημερομηνία. Στις 5 να τους πάτε στα δικαστήρια, να τους τραβήξετε στα δικαστήρια. Στις 5 Δεκεμβρίου. Αν δεν το κάνετε εσείς θα το κάνω εγώ. γιατί αλλιώς ε, τίποτα δεν πρόκειται να κάνουν Θέλω να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά, σύντομη θα είμαι, αλλά εκτός μικροφώνου δεν ακούγεται η ομιλήτρια. Στη Λεμεσό θα είναι υπουργό Μεταφορών. Εγώ ήθελα μόνο να σας πω ότι υπάρχει ομοφωνία στην προκειμένη περίπτωση. Σα υποστηρίζουμε. Πρέπει να κάνει κάτι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Προσπαθεί να επιβάλλει το Συμβούλιο. Τι κάνατε, αντιγράψατε απόσπασμα από την ομιλία μου. Σαν κροκόδηλος είναι το Συμβούλιο έρπεται και κολυμπάει κάτω από την επιφάνεια του νερού και ε, ξαφνικά επιτίθεται όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Είναι δόλιο το Συμβούλιο, σας το λέω έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, ε, πριν ακούσουμε τον Τζούτζ και πάλι και περάσουμε και στο θέμα του κυρίου Γκρίφιθ, τι έχετε να μας πείτε. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους, θα είμαι σύντομος. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαζεμπόσκι, εξαιρετική η εργασία του. Ε, ήταν μακρά η περίοδος της αξιολόγησης και τώρα φτάσαμε στο πέρας ε, της διαδικασίας αξιολόγησης. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σα ότι πρέπει να περατωθεί η διαδικασία. Η πρόθεση της Επιτροπής είναι αυτό ακριβώς να κάνουμε, διαδικασία επί παραβάση. Αλλά είναι χρονοβόρα η διαδικασία και δυσχερής. Πρέπει να είναι παρκώ στοιχειοθετημένη η υπόθεση από νομική πλευράς για να τα καταφέρουμε. Ε, αυτό το ζήτημα της Λεμεσού θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση εκ παραλίλου. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη στο μέτρο το δυνατό για να έχουμε απτά αποτελέσματα, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια που εξακολουθούν να ε, υπάρχουν λόγω μίας και μόνο λέξης, δύο μάλλον στα ελληνικά, εθνική κυριαρχία. Είναι δυσεπίλητο το ζήτημα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Οπότε όλοι αυτοί έχουν υπογράψει. Εσεί, μου λέτε και ξανά, μου λέτε για κυριαρχία. Μα το υπέγραψαν, το συμφώνησαν. Υπέγραψαν και κόντρα υπέγραψαν. Δηλαδή, τι, τι, τι να χρησιμοποιήσουν ω δικαιολογία. Έχουν συμμογράψει μια νομική συμφωνία και ναι, ξέρω, λέτε ότι παίρνει χρόνο κτλ. αλλά ακόμη περισσότερο θα πάρει άμα δεν ξεκινήσουμε στι 5 Δεκεμβρίου. Ε, πρέπει αυτούς τους, ε, τα κράτη-μέλη να τα επιφέρει στην τάξη. Δηλαδή να δουν αυτά που έχουν υπογράψει. Έχουμε ένα σύστημα όπου όλοι πρέπει να υπακούν τους νόμους εκτός από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ε, δεν είναι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Τζόρτζο. Ευχαριστώ πολύ για την ιδέα αυτή που έχετε για παράταση αυτή τη εντολή. Είναι καλή ιδέα, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει. Εγώ ευχαρίστω. Γιατί ε, δεν μου αρέσει να τα αφήνω στη μέση τα πράγματα. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ. Και εδώ νομίζω είμαστε σε, στο ίδιο μήκο κύματο. Πρέπει να αρχίσουμε τη διαδικασία κατά παράβαση όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν είναι πολύ εύκολα. Ε, όμως Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Επίσης, είμαι κατά του να λέμε πολλά λόγια σε σχέση με το SES3, γιατί κάποιες χώρες μπορεί να περιμένουν το SES3 για να δουν ποιο είναι το καλύτερο. Ναι. Αυτό είπα στην ομιλία μου ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες πρωτοβουλίες. Και αυτά που είπατε κάποια από εσά είναι πολύ σημαντικά ότι δηλαδή ένα από τα βασικά προβλήματα για τη διοργάνωση της συνεργασίας η, η ολοκλήρωση του SES στο NSP είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες για την απασχόληση της συντάξης, τις μεταφορές από τη μια εταιρεία στην άλλη. Από αυτή την άποψη μπορεί κανείς να σκεφτεί κάποιες πρωτοβουλίες. Η Υπουργοί Μεταφορών, να σας πω κάτι, δεν το παίρνουν στα σοβαρά το θέμα. Δεν ε, θέτουν τα πολιτικά ερωτήματα, δεν το αντιμετωπίζουν. Φοβούνται. Φοβούνται τη, τα συμφέροντα των θεσμών και των απασχολούμενων εκεί. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αν κανείς τώρα κοιτάξει την ΦΑΜΠΕΚ, για παράδειγμα, ένα ε, χώρος είναι, ένα αέριο χώρος. Άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά άκουσα πως υπήρχε μια προσπάθεια ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές χώρες να ε, πετούν στη, σε πιο στενή, στη πιο ευθεία γραμμή. Μετά όμως είπαν οι εταιρείε ότι άμα στην ευθεία γραμμή εγώ χάνω χρήματα. Ε, άρα δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Κάποιο ASP ε, δεν θέλει να χάσει έσοδα και θα μας κάνει βόλτες και γύρες πάνω στον ουρανό. Πολιτική βούληση λοιπόν από τους υπουργούς, αλλά και σε όλα τα επίπεδα, κρατικό, NSP και NSA, χρειαζόμαστε ένα κοινό πνεύμα. Θέλουμε να δουλέψει αυτό το πράγμα, θέλουμε να το καταφέρουμε και αυτό το έχουμε χάσει. Για να επανέλθω στο ΦΑΜΠΕΚ, για τον εναέριο χώρο δεν είμαι βέβαιος, για να είμαι για τα στρατικά θέματα για την ώρα, αλλά πιστεύω πως μπορούν να βελτιωθούν ακόμα πολλά. Το κύριο, ερώτημα όμως είναι πώς φτιάχνουμε οδικό χάρτη Πώς φτιάχνουμε οδικό χάρτη. Οι Γάλλοι θέλουν να το φτιάξουν ένα κρατικό όμιλο διοικητικών οργανισμών, ενώ άλλοι θέλουν ιδιωτικό. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και δεν έχει λυθεί εδώ και δύο χρόνια και πάνε από το Μάταχα στο Λόβεν και οποιαδήποτε άλλη πόλη. Πολλοί κοντέψαν, κοντέψαν το Σεπτέμβριο να σκεφτούν τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας, μεικτής εταιρεία ε, ε, για αρχή. Τι θα έπρεπε να είναι Φερχάιν, που όπως λέμε στα γερμανικά, ανώνυμος εταιρεία, στα γαλλικά, ε, Société Anonyme. Δεν μπορούσαν καν να συμφωνήσουν για το καθεστώς εταιρεία. Φτου και πάλι αναβολή. Δηλαδή, πολιτική βούληση από πλευρά των Υπουργών είναι ανύπαρκτη. Κάποιοι Υπουργοί, για να μην πω τι χώρε του, Είπε ο Υφυπουργό ότι το δικό μου Εθνικό Υπουργείο είναι τόσο ισχυρό που δεν θέλω εγώ να τώρα να μπλεχτώ. Οι άλλοι είπαν ότι αν θέλουμε κάτι να αλλάξει, ε, ε, μάλλον αν κάνουμε πως αλλάζουμε κάτι θα κατέβουν σε απεργία. Και δεν θέλω αυτό να το ρισκάρω γιατί ο Πρωθυπουργό μου θα με σκοτώσει έτσι και γίνει απεργία. Και δεν κινούνται. Είναι θέμα πολιτικού θάρρους και αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε, να πάρουμε, να τραβήξουμε μαζί μας και τους απασχολούμενους, τους εργαζόμενους. Έχουμε εμπειρία. Υπάρχουν παραδείγματα όπου στο ΦΑΜΠ ε, τραβούν, προσελκύουν τους εργαζόμενους με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ σε άλλα FAB δεν τους μιλάνε καν στους εργαζόμενους και είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι θα εμποδίσουν οποιαδήποτε αλλαγή, κίνηση κτλ. γιατί φοβούνται μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό το είδος η συνεργασία ανάμεσα στα Υπουργεία, τις οργανώσεις και τα συνδικάτα δεν υπάρχει. Μα δεν είναι τελείως κατά τα συνδικάτα, δεν είναι και υπέρα, αλλά σίγουρα δεν είναι απόλυτα κατά. Αν βρούμε δικούς χάρτες συνεργασίας και τα λοιπά, θα είναι ο καλύτερος τρόπος. Και τώρα για το ΦΑΜΠΕΚ, τα ε, πω απλά γιατί ο Πίτερ με κοιτάει στραβά. Ε, εκεί έχουμε μια κατάσταση όπου το FAPC ε, όπου κάποιες χώρες έχουν πάρα πολύ προσωπικό στο, στα κέντρα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας ενώ άλλες δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Πώς τα οργανώνουμε αυτά. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, γιατί είναι θέμα χωρητικότητας και αποτελε... Ε, κόστους τα κτλ. Πρέπει να βρεθεί λύση και εδώ χρειάζεται πίεση. Για να δω τι άλλο ξέχασα. Νομίζω πως μπας περιπτώσει πήρατε το μήνυμα για την FABEC. Έχουμε πρόβλημα με την MUAC. Με το MUAC που είναι ένα πολύ καλό σύστημα. Είναι το κέντρο ελέγχων και κυκλοφορίας του Μάστριχτ είναι, η Γαλλία και η Ελβετία σκέφτονται ακόμα αν θα μπουν σε αυτό το κέντρο ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας. Το θέμα είναι, είναι ένα κέντρο τέτοιο ή είναι ένα κέντρο κρατικό ANSP. Ε, ε, ε σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ για την, τις ερωτήσεις σας. Υπάρχουν τρόποι να επανέλθουμε. Διάβασα την έκθεση αυτή για το τι σημαίνει στη χώρα μου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. George, thank you very much. Right now... Ευχαριστούμε, George. Ο κύριος Γκρίφιτς από το Σώμα Εξέτασης της Απόδοσης. Άμα κανείς δεν κάνει τίποτα, πώς μπορεί να κάνετε έκθεση για την απόδοσή του. Φαντάζομαι θα μας φωτίσετε. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ευχαρίστω να έρθω εδώ να σας μιλήσω για, σε ένα σώμα το οποίο είναι υπέρ του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και μεγάλη μου χαρά να κάθομαι μαζί με τον κύριο Γερζεμπόφσκι. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια θέματα κλειδιά. Όταν σας μίλησα την περασμένη φορά, θέλατε να γνωρίζετε ποια ήταν η πρόοδος για την εξέλιξη του σχεδίου Εξέταση της προόδου και με χαρά μου μπορώ να σας πω ότι τα 29 σχέδια για τα οποία έπρεπε εμείς να κάνουμε αναφορές έχουν εισέλθει. Δεν έχουν πετύχει τους στόχους, αυτό είναι σαφές. Λίγο έχουν πέσει έξω, αλλά δεν έχουν επιτύχει τους στόχους πάντως. Είναι μείωση σε σχέση με τα όσα είχαμε αρχικά προβλέψει να κάνουμε στην πρώτη έκθεση που είχε εκπονηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 2010 και που ήταν πολύ πιο φιλόδοξη. Ε, είδαμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να ε, μειώνουν τις φιλοδοξίες τους σε μεγάλο βαθμό και αυτό ταιριάζει και με τα όσα είπε ο Τζόρτζ. Εμείς περιμέναμε διαρθρωτικές αλλαγές να ξεκινήσουν στο πρώτο ΑΡΠΗ ώστε μέχρι να φτάσουμε στο σχεδιασμό του δεύτερου αρπή να είχαμε ήδη κάποια ωφέλη που θα είχαν αρχίσει να διαφαίνονται δεν φαίνονται ωφέλη. Ε, ακούσαμε και από τον Τζόρτζ ότι υπάρχουν τα σχέδια απόδοσης των ΦΑΠ και τη συμβολή αυτής της απόδοσης. Ε, δεν θα σας εκπλήξει να σας πω ότι δεν υπάρχει απόδοση ε, μέχρι στιγμής. Και έτσι ερχόμαστε σε, αυτό, ε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Παρακολουθούμε τα κράτη, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα παρακολούθησης και μετά από αυτή τη βδομάδα λοιπόν, θα κλείσουμε τη διαδικασία επικύρωσης θα αρχίσουμε να απελευθερώνουμε κάποιες πληροφορίες ώστε να δείτε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Αργότερα αυτή τη βδομάδα λοιπόν θα δείτε τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση πρόοδου. Αυτό που έχει επίση συμβεί είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ότι δηλαδή κατά πόσο θα πάμε στα δικαστήρια για όσα πράγματα δεν λειτουργούν. Η Κομισιόν έχει ήδη προβεί σε δράση για λογαριασμό μας και το σύστημα είναι πολύ αποτελεσματικό, αρχίζει να λειτουργεί. Η στήριξη που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετική. Τώρα ξεκινάμε με μια πολύ σπουδαία δουλειά και εδώ ίσως τα κράτη-μέλη να πρέπει να παίξουν πια το ρόλο τους, γιατί στη δεύτερη περίοδο αναφοράς που αρχίζει το 2015 πρέπει να αρχίσουν να προσχεδιάζουν από τώρα. Μέχρι τα τέλη του έτους αναμένουμε λοιπόν τις συμβολές των κρατών. Ε, ιδιαίτερα τρία κράτη που δεν συνέβαλαν την περασμένη φορά, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Περιμένουμε να κάνουν επιπλέον προσπάθειες αυτοί και τους το έχουμε καταστήσει σαφές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης σε σχέση με τις ε, περιόδους αναφοράς. Ότι δηλαδή αυτή τη φορά δεν προσπάθησαν, οπότε αναμένουμε την επόμενη να κάνουν κάτι την επόμενη περίοδο, περίοδο σχεδιασμού. Έχουμε μια βασική, ένα βασικό σενάριο, ένα σενάριο που όλοι αναγνωρίζουμε καθημερινά, δηλαδή το μήνυμο που θα μπορούσαν να επιτύχουν αν έμεναν με τα πράγματα όπως έχουν. Και έπειτα να δούμε και τη διαρθωτική αλλαγή και ακούγοντας τα όσα είπατε πριν από λίγο είναι ότι χρειάζεται αυτή η διαρθωτική μετακίνηση ώστε να έχουμε τα ωφέλη. Θα σχεδιάσουμε λοιπόν το τι θα συμβεί αν έχουμε όλες τις διαρθωτικές αλλαγές που θέλουμε για να φτιάξουμε στόχους που θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Επίσης ε, έχουμε ένα σενάριο μέσα στο πλαίσιο του πακέτου ΣΕΖΑΡ. Έχω γράψει τον επικεφαλή του προγράμματο ΣΕΖΑΡ, ζητώντα του να μου δώσει το υλικό που χρειάζομαι μέχρι τι 7 Δεκεμβρίου για να κάνω αυτό το διαδικασία σχεδιασμού. Οπότε έχουμε μια ιδέα για το τι θα αποδώσει το ΣΕΖΑΡ μέχρι τότε. Τέλος, σε στρατιωτική και τεχνολογική αλλαγή, αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά που θα είναι το άλλο σενάριο, το εξαιρετικά φιλόδοξο. Αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και συμπληρώνονται από μια εργασία που είναι το RP2 γεγονές και οι συμβουλές προς την Κομισιόν τις έχουμε ήδη δώσει στην Κομισιόν και περιμένουμε να μας δώσουν τη δική τους άποψη. Είναι πολύ θετικά λοιπόν όλα αυτά. Έχει υπάρξει πρόοδος, υπάρχει μεγάλη, πολύ σπουδαία σχέση ανάμεσα σε τον Ζόρτζο Γερζιμπόφσκι και σε μένα. Ε, συζητάμε πάντα για το τι μπορούμε να επιτύχουμε. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα από όσα κάνουμε μέχρι στιγμής για να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, ε, σχόλια. Εγώ έχω μια ερώτηση. Μπορεί να σας ε, φαίνεται αυτονόητο και ηλίθιο, αλλά θα το ρωτήσω παρόλα αυτά. Γιατί δεν έχουν τις ευκταίες επιδόσεις τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Εσείς ε, κάνατε τη σύνοψη των σημείων που αιτιολογούν τις κακές επιδόσεις. Δεν ασκείται επαρκή πίεση. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι χρειάζεται πολύ καλύτερες επιδόσεις. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το πρότυπο που χρησιμοποιούμε, δηλαδή η διαφορά στην ε, ε, τιμολόγηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τη ΣΥΠΑ έχουμε μία βάση 100 ευρώ. Αν τώρα ε, κάνουν αυτά που είπαμε θα κάνουν, θα φτάσουμε στα 690. Καταλαβαίνετε πόση απόσταση μας χωρίζει από αυτό το στόχο. Ε, ταυτόχρονα μειώνεται η εναέρια κυκλοφορία. Πρέπει να σας πω όμως, Πρόεδρε, ότι δεν πρόκειται μόνο για τις εθνικές αρχές που δεν συμμορφώνονται, αλλά είναι και οι ίδιοι οι αερομεταφορείς Δηλαδή του γνωστοποιούνται ότι υπάρχουν εναλλακτικέ οδοί, αεροπλοίες και δεν τι χρησιμοποιούν όμω. Οπότε θα πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσερ στο Κέσσερ. Ναι, λέει ο πρόεδρο, αλλά το βασικ... η βασική τροχοπέδη είναι η έλλειψη πολιτική βούληση όμω. Ε, για να δούμε αν έχει κάτι να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είστε και υποχρεωμένος, αλλά να έχετε τη δυνατότητα τουλάχιστον άμα θέλετε. Ναι, Πρόεδρε, εν συντομία για να επιβεβαιώσω αυτά που μόλις μας είπε ο Πίτερ. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με τον Οργανισμό Αναθεώρησης ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με, ε, με τον προγραμματισμό για τις επιδόσεις τους και τον προσδιορισμό των κανόνων του παιχνιδιού για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς. Ε, πρέπει να αντιληφθείτε ότι οι επιδόσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της πρωτοβουλίας ΣΕΣΕ και παρότι τα ΦΑΠΣΕ, οι διαχειριστές των δικτύων, το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ καλύπτουν το θέμα της επίδοσης πρέπει να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα διότι έχει μεγάλη σημασία και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και εγκαίρως. George, να υπενθυμίσω κάτι που είπα για τις νέες πρωτοβουλίες που μπορούμε να εξετάσουμε. Ένα από τα τελευταία παραδείγματα ήταν το πώς μπορούμε να καταστήσουμε δεσμευτικούς τους στόχους περί επιδόσεων, γιατί προς το παρόν η νομοθεσία σε δεν ε, περιέχει δεσμευτικούς στόχους. Μπορεί να κάνει απλώς ε, σχόλια και συστάσεις η Επιτροπή για να θεώρηση των στόχων. Αν όμως δεν θέλουν, όπως εξάλλου έγινε και από τρεις μεγάλες χώρες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξού και το ζήτημα. Πώς, ε, με ποιο τρόπο να καταστήσουμε δεσμευτικούς τους στόχους. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Πρόεδρος, δίκιο έχεις, Τζόρτζ, αλλά ε, από την ε, εμπειρία που έχω μέχρι στιγμής από το Συμβούλιο δεν έχει καμία σχέση, είτε είναι δεσμευτική είτε όχι οι στόχοι, ό,τι θέλουν κάνουν. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Κύριε Γκρίφιθ, μου θυμήσατε και κάτι άλλο και θα ρωτήσω το εξή. Τι αερομεταφορές δεν χρησιμοποιούν τις εναλλακτικέ ε, οδούς, διαδρομές. Ε, τι κάνετε, προσπαθείτε τώρα να μου καταστρέψετε την ομιλία της Πέμπτης, αναφερόμουν σε αυτό το ή άλλως. Ε, πρόκειται για μια υπηρεσία που συνδιαχειρίζεται το Άμστερνταμ και το Μιλάνο. Mm. Ε, και για τις εναλλακτικέ ε, διαδρομές ε, το πρόβλημα είναι ότι οι αερομεταφορείς δεν έχουν το απαραίτητο λογισμικό για τον προγραμματισμό των πτήσεων. Οι μεγάλοι αερομεταφορείς έχουν λογισμικά που είναι συμβατά με αυτό του Eurocontrol. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε συνολικά το πακέτο ΣΕΣ για την πρόθεση των επιδόσεων. Είτε μιλάμε για τους διαχειριστές δικτύου, είτε για τις, ε, τα λειτουργικά ε, τμήματα ε, εναερίου χώρου. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πρώτον ότι γνωρίζουν τις εναλλακτικέ διαδρομές οι αερομεταφορές, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ο διαχειριστής δικτύου έχει την εξουσία, παραδείγματο χάρη, να ζητήσει από κάποιον αερομεταφορέα υποχρεωτικά να αλλάξει τη διαδρομή του. Ε, πρόεδρος, αφού δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα κάνω εγώ και άλλη μία. Σχετίζεται αυτό με τους Αμερικανούς ε, και την επόμενη σύσκεψη. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης ε, και ε, παρακολουθούμε αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί όπως εκείνοι ε, που ε, παρακολουθούν αυτά που κάνουμε εμείς. Το βασικό ζήτημα αξιολόγησης ποιο είναι του χρόνου αναμένεται αναθεώρηση του συστήματος και θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι διαφορές ανάμεσα ανάμεσα στα δύο συστήματα. Καλά, ούτως ή άλλως ε, είναι μεγάλο κεφάλαιο Αμερικανή, λέει ο Πρόεδρος. Θα τα αφήσουμε άλλο Παπαευαγγέλιο, Ευαγγέλιο αυτό. αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε και τους δύο που ήρθατε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε με τις ε, παρούσες ιδιότητές σας ε, στο... για την μελλοντική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Ίσως πιούμε και καμιά μπυρίτσα στη Λεμεσό. Γιατί μπορεί να ακούσατε ότι μπορεί να χρειαστώ και προσωπική προστασία, security στη Λεμεσό από αυτά που θα πω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Μέση διάταξη. Να σα υπενθυμίσω μόνο ότι τη Δευτέρα στις 5 Νοεμβρίου, 3 το απόγευμα στις Βρυξέλλες ε, θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση και έχουμε τη μεγάλη και σημαντική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, αλλά στις 6 Νοεμβρίου. Να ευχαριστήσω τους πολισταμένους και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, λύεται η συνεδρίαση.